Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. Παρακαλώ καθίστε. And we can begin our meeting. Να ξεκινήσει η συνεδρίαση. we begin already? Yeah. All right. I open the meeting of the... Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ενημερώσω πως θα απουσιάζουν δύο συνάδελφοι, μας ενημέρωσαν. Η κυρία Βάνα, σε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γυναικών στη Νέα Υόρκη. Και ο κ. Ντόιτς έχει ανηλυμένη υποχρέωση στην περιφέρειά του στην Ουγγάρια. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Γιατί είναι εδώ. Αύριο, αύριο. Α, είναι εδώ ο κύριος Ντόιτς. Δεν θα είναι αύριο εδώ, μάλιστα. Γι' αυτό άλλαξε η μερίσια διάταξη. Και να σας ενημερώσω λοιπόν για την αλλαγή αυτή, γιατί κύριος Ντόιτς, λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεων που είπαμε, ζήτησε η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης του να αναβληθεί για τις συνεδρίες του Απριλίου. Οπότε, με τις αλλαγές αυτές ε, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη, ναι, έτσι νομίζω. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 15 και 16 Φεβρουαρίου. Τα σχέδιο πρακτικών είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για να σώσουμε κανένα δέντρο. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ε, μέχρι το τέλος συνεδρίασης τα πρακτικά εγκρίνονται. Ωραία, δεν υπάρχει σχόλιο. Δεν έχω κάποια άλλη ανακοίνωση. Και άρα ξεκινάμε με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ένα εργαστήριο, ας πούμε, για την απλοποίηση της ε, πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας μετά από συνεδρίαση στις 15 Οκτωβρίου και το ψήφισμα πέρσι τον Νοέμβριο και μετά από την ανταλλαγή απόψεων με την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση του κυρίου Κάλασα ε, σήμερα θα ξαναδούμε το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας ζήτησε από τη μονάδα έρευνας ε, που υποστηρίζει το έργο μας να οργανώσει ένα εργαστήριο για την απλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Όπως βλέπετε στο πρόγραμμα θα ακούσουμε αρκετούς ειδικού ε, επί του θέματος. Θα κάνω μια εισαγωγή και αφού ακούσουμε τους ειδικού μας θα ακούσουμε και τους βουλευτές. αλλά και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Έχουμε επίσης κάποιους ε, προσκεκλημένους από την Επιτροπή των Περιφερειών και θα ήθελα να ακούσω την άποψή τους γιατί η Επιτροπή των ε, Περιφερειών ε, οργανώνει και εκείνη κάποιες σχετικές εκδηλώσεις. Οπότε η απλοποίηση της πολιτικής συνοχής θα είναι πάντα κάτι το οποίο ανησυχούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας, ειδικά όσον αφορά τους δικαιούχους. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της απόδοσης της πολιτικής ε, συνοχής και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η μείωση του διοικητικού βάρους ε, επί των δικαιούχων και των διαχειριστικών φορέων επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και μειώνει και τον κίνδυνο λάθος. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το 2014 μέχρι το 2020 μας δίνει δυνατότητες μείωσης του διοικητικού βάρους και να απλοποιηθεί η πρόσβασή τους ε, στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Παρόλες τις ε, προσπάθειες φαίνεται πως ε, πάρα πολλές διαχειριστικές αρχές θεωρούν πως η πολιτική συνοχή έχει γίνει πιο γραφειοκρατική και χρονοβόρος το θέμα αυτό έχει απασχολήσει όλα τα θεσμικά όργανα και είχαμε ήδη αναλάβει δράση το 2015 για να δούμε ποιες είναι οι ρυθμιστικές επιλογές που έχουμε όσον αφορά την απλοποίηση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ε, η πολυπλοκότητα αυτού του ζητήματος ε, εν μέρη βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία. Σε μεγάλο βαθμό δεν βασίζεται σε κανόνες που υπάρχουν και σε άλλους τομείς όπως η πολιτική του ανταγωνισμού οι οποίοι όμως συχνά δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες. Το ψήφισμα του Νοεμβρίου 2015 που εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε τη σημασία της περαιτέρω απλοποίησης της πολιτικής συνοχής και τόνισε το ότι η εφαρμογή, η διαχείριση, οι αναφορές ε, και ο έλεγχος ε, των ε, ταμείων αυτών εξακολουθούν να είναι μηχανισμοί δυσκίνητοι και για τους δικαιούχους και για τις διαχειριστικές αρχές ειδικά για όσους δεν έχουν τόσο μεγάλες διοικητικές δυνατότητες. Έτσι ζητήσαμε από το Τμήμα Πολιτικής να κάνει κάποια έρευνα και σήμερα έχουμε μια πρώτη τέτοια συνεισφορά στην Επιτροπή μας. Θα εστιάσουμε λοιπόν στα εξής ε, θέματα. Την ηλεκτρονική συνοχή, απλοποιημένο κόστος, ε, κανόνες ελέγχου ανάλογα με τα κράτη-μέλη και τις διαχειριστικές αρχές και βεβαίω ε, θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Οπότε Αυτά τα ολίγα ως εισαγωγή από εμένα. Έχουμε λοιπόν συνήθως ε, λίγο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι και να μην μιλήσετε για περισσότερα από 8 λεπτά σε κάθε παρουσίαση για να σας ακούσουμε όλους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπως αυστηροί για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους ε, συμμετέχοντες. Θα ξεκινήσω δίνοντας τον λόγο στον κύριο Ρόναλντ Μπλούμερ, διευθυντή της Blue Sons, ο οποίος θα μας μιλήσει για την, ε, τις απλοποιημένες επιλογές ε, κόστους ε, στην πράξη. Λοιπόν, έχετε τον λόγο και θα ακούσουμε και τους άλλους ομιλητές. To... ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαήλου που θα προσπαθήσω να μείνω στα στενά χρονικά όρια που μου δώσατε. Κατά βάση θα ήθελα να σας παρουσιάσω την μελέτη που μας ζήτησε να διεξαγάγουμε το τμήμα Β και δρομολογήθηκε το Δεκέμβριο η διενέργεια της μελέτης αυτής. Θα σας πω καταρχάς ε, λίγο σύντομα ποια είναι η δομή της παρουσίασης. Θα σας παρουσιάσω τη μελέτη καταρχάς και θα σας πω σίγουρα πράγματα που γνωρίζετε, ποιες είναι αυτές οι απλοποιημένες επιλογές κόστους και θα σας αναφέρω και τα πρώτα πορίσματα της μελέτης. Πολύ γρήγορα λοιπόν, τι προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα είναι η χρήση ε, των απλουστευμένων αυτών επιλογών από τα διαφορά κράτη-μέλη και αυτό σε δύο περίοδους προγραμματισμού, δηλαδή 7 13 και 14 έως 20. Όπως σας είπα, ξεκίνησε η μελέτη το Δεκέμβριο και θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας μέσα Απριλίου του τρέχοντος. Βασιστήκαμε και σε μελέτη βιβλιογραφίας και εκεί που πιστεύω ότι μπορεί να ε, συνιστά η μελέτη μας προστιθέμενη αξία σε έρευνα της Κομισιόν, της Γαμαδέλτα ΡΕΓΙΟ και Employment, αυτό που κάναμε είναι ότι ακούσαμε τις διαχειριστικές αρχές, τους δικαιούχους ε, από τα διάφορα κράτη-μέλη για να δούμε ποια είναι η δική τους εμπειρία είτε κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού είτε κατά τη νέα περίοδο που μόλις ξεκίνησε. Έχω βάλει και κάποιες σημαίες κρατών μελών για να δείτε ποια είναι τα κράτη-μέλη που ακούμε. Γενικά έχουμε επαφέ με διάφορους εμπλεκομένους φορείς και θέλουμε να συλλέξουμε ε, το feedback από όλους αυτούς. Η κυρία Μιχαήλοβα αναφέρθηκε στους στόχους πάντα στο πλαίσιο της απλούστευσης θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα του πλαισίου των διαρθρωτικών αυτών ταμείων και εσείς είπατε ότι στόχος είναι ε, μείωση διοικητικού άκθους όπως προείπα εγώ και μακροπρόθεσμα, δηλαδή στόχος είναι η πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων εστιάζοντας περισσότερο στο περιεχόμενο στους στόχους, πολιτικές και όχι τόσο στο διαχείριση και στον έλεγχο Υπάρχει και ένα ιστορικό ε, πίσω από τους τρεις βασικούς τύπους ε, των επιλογών μας. Ξεκινήσαμε στην τελευταία περίοδο προγραμματισμού το 2006 για το Κοινωνικό Ταμείο αρχικά, μετά κάλυψε και το ΕΤΠΑ ε, και με μια τροποποίηση του 2010, νομίζω τότε 15 κράτη-μέλη χρησιμοποιούσαν τις απλοποιημένες επιλογές κόστους στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κάτι που σίγουρα γνωρίζετε, τρεις είναι οι βασικοί τύποι ε, που μας απασχόλησαν ε, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Πρώτα απ' όλα οι λεγόμενοι πάγοι συντελεστές, δηλαδή πώς μπορούμε να αποφύγουμε να συλλέγουμε όλα τα εισιτήρια και όλες τις αποδείξεις και τιμολόγια. Έχουμε λοιπόν μηχανισμό εδώ που η δήλωση του έμεσου κόστους ε, γίνεται με βάση ένα ποσοστό του άμεσου κόστους ε, και βέβαια δεν απαιτούνται πλέον ε, τα αποδεικτικά έγγραφα, τα δικαιολογητικά για τα έμεσα έξοδα, μόνο για τα άμεσα. Δεύτερο, ο κόστος, ε, εδώ η επιστροφή του κόστους γίνεται με βάση καθορισμένες μονάδες κόστους, ώρες κατάρτιση και τα λοιπά, όλα αυτά μπορούν να τυποποιηθούν και η επιστροφή ε, εξαρτάται από τον αριθμό των μονάδων ε, κάστοτε. και τέλος η καταποκοπήν, τα καταποκοπήν ποσά, δηλαδή έχουμε ένα προκαθορισμένο κατά αποκοπήν ποσό για μικρά project και η πληρωμή γίνεται με βάση την εκτέλεση δραστηριότητας. Βλέπουμε λοιπόν και τη χρήση, βλέπουμε και την εμπειρία, ποια είναι τα πρώτα πορίσματα. Θέλουμε να δούμε άμεσα οι στόχοι πώς επιτεύχθηκαν, βοηθά δηλαδή ε, το απλοποιημένο κόστος, τη μείωση του διοικητικού άχθους και τελικά σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται και οι πιο ευρύ στόχοι που προανέφερα, δηλαδή η επανεστίαση των πόρων ε, στους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής, δηλαδή περισσότερο να ασχολούμαστε με την εφαρμογή και την συνέχεια και όχι με τον έλεγχο και την επαλήθευση και τέλος ε, κάποιες από τις δυσκολίες ε, που μας ανέφεραν οι περιφέρειες και τα κράτη κατά την εισαγωγή χρήση αυτών των οπλιστευμένων επιλογών είναι το τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, των οπλιστευμένων αυτών επιλογών, μέχρι στιγμής δεν έχουμε συστηματικά δεδομένα για το ε, ΕΤΠΑ. Έχουμε καταρχήν κάποια στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που μας βοηθούν κάπως να καταλάβουμε και την χρήση σήμερα αλλά και ε, τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι επιλογές. Γύρω στο 7% ε, του έκτα δηλώθηκε στο πλαίσιο των αυτευμένων ε, επιλογών το, την περίοδο 7-13 και είχαμε και μια έρευνα της Δέλτα απασχόλησης που δείχνει αύξηση για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Το ποσοστό το αντίστοιχο λοιπόν γύρω στο 35%. Δεν έχουμε όμως συστηματικά δεδομένα όπως είπα. Δεν έχουμε στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφέρειας Ανάπτυξη. Ελπίζουμε να διατεθούν ε, σύντομα η ΓΔ Ρέγγιο έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να καταγραφούν αυτά τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά το feedback, γιατί ε, χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη ε, περισσότερο αυτά, αυτές τις επιλογές και πώς εξηγείται αυτή η άξη του ποσοστού Πρώτα απ' όλα έχουμε μεγαλύτερη του ρυθμιστικού πλαισίου, δηλαδή υπάρχει πλέον η πεποίθηση ότι είναι, μεγάλη, είναι πολύ καλύτερη ποιότητα και για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιλογές υπάρχει καθοδήγηση, ενημέρωση και αυτό έγινε και σε πιο πρώιμο στάδιο, νωρίτερα δηλαδή στο στάδιο της μελέτης, του σχεδιασμού των προγραμμάτων. Άρα οι απλουστευμένες επιλογές τελικά φαίνεται να επιτυγχάνουν τον άμεσο στόχο της μείωσης του διοικητικού άχθους. Παραλαμβάνω ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά, πρέπει να μιλήσουμε και με τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι από τις συνεντεύξεις που είχαμε. Είδαμε ότι υπάρχουν θετικές προσδοκίες ότι αφορά τη μείωση των απαιτήσεων ε, στη φάση της ε, αναφοράς ε, και της πληρωμής αλλά βέβαια και της υποβολής του προγράμματος και στην περίοδο 14-20 με τη χρήση των επιλογών αυτών που είναι περιορισμένη βέβαια γιατί πολλά project δεν έχουν παρκώς προχωρήσει για να φτάσουν σε αυτή τη φάση δηλαδή στη φάση της πληρωμής ή επιστροφής δαπανών αλλά θα δούμε στη συνέχεια πιστεύουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θετικό ήταν και το feedback σε σχέση με κάτι που ανέφερε η κυρία Μιχαήλουβα, δηλαδή τη μείωση των ε, ποσοστών σφάλματος το ελεγκτικό για την πρώτη περίοδο ε, δημοσίευσε κάποια απορίσματα και δείχνουν μείωση των ε, ποσοστών λάθους. Αυτά θα ε, βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Επίσης, προσέλκυση νέων ετούντων. Εδώ είναι κάπως συγκεχημένο το αποτέλεσμα. Ναι, μεν μειώνεται η πολυπλοκότητα, διευκολύνεται το έργο και των πιο μικρών ετούντων που δεν έχουν μεγάλες ομάδες για τη διαχείριση, αλλά ε, σε κάποιες περιφέρειες ε, μας είπαν ναι, έχουμε νέους σε άλλες περιφέρειες όμως ε, δεν θεώρησαν ότι υπήρξαν αρκετά κίνητρα για κάτι τέτοιο. Τώρα, ευρύτερη στόχη, δηλαδή όχι μόνο μείωση του διοικητικού άκου, αλλά κάτι που επίσης αναμένεται είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη εστίαση και επικέντρωση στους στόχους της συνοχής, όπως είπα, στην εφαρμογή, το follow-up και εδώ έχουμε θετικό feedback ε, σε σχέση με το ότι παραδείγματος χάρη χρειάζεται λιγότερος χρόνος ε, για τον έλεγχο, αλλά δεν έχουμε ακόμη αποδεικτικά στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι ε, αυτό σημαίνει ότι αφιερώνεται περισσότερο χρόνο στην εφαρμογή. Εύκολο να καταλάβει κανείς το λόγο γιατί είναι διαφορετικά τα άτομα που είναι αρμόδια για παράδειγμα για τον χρηματοοικονομικό έλεγχο δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ε, εφαρμογή. Βλέπουμε από κάποιες περιφέρειες μάλιστα να ε, μειώνεται το προσωπικό. Ε, δηλαδή να μην στελεχώνεται περισσότερα άτομα για την εφαρμογή. Για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα, όπως είπα, υπήρξε σημαντική αύξηση μένα. υπάρχουν όμως και δυσκολίες με την εισαγωγή και τη χρήση αυτών των επιλογών. Αυτά τα δεδομένα που βλέπετε είναι από τη Δέλτα απασχόληση, μια έρευνα για τη χρήση ε, αυτών των επιλογών. Βλέπετε ότι είναι σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη δηλώνουν το πραγματικό κόστος, αυτό όμως αποτελεί πια εξαίρεση. Λουξεμβούργο, Σουηδία, άλλα μέλη, Ιταλία, σημαντικοί ε, χρήστες των απλουστευμένων επιλογών. Άλλα κράτη-μέλη όμως, Βουλγαρία, επί παραδείγματι, Ουγγαρία, Γερμανία. Εδώ βλέπουμε μέτρια χρήση των αποστευμένων επιλογών κόστος. Ποιο είναι το feedback που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν ε, στο στάδιο της εισαγωγή αυτών των ε, επιλογών. Έγινε πολλή συζήτηση ότι αφορά ε, το ότι δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή δεν νιώθουν σίγουρα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιλογές. Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιο σαφές αυτό είναι σίγουρο, αλλά υπάρχει ακόμη ο φόβος ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια ερμηνεών και επειδή δεν υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση, υπάρχουν διαφορετικέ μέθοδοι για τη χρήση των ε, επιλογών και υπάρχει ο φόβος ότι όταν αργότερα έλθουν οι ελεγκτές να μην θεωρήσουν έγκυρη την επιλογή σαν μέθοδο και να μην επιστραφούν τα ποσά. Υπάρχουν ε, θέματα επίσης ε, ασυμβατότητας με την εθνική περιφερειακή σε κάποια κράτη νομοθεσία όπου χρειάστηκε μάλιστα να αλλάξουν ε, τα εθνικά ή ε, περιφερειακά ρυθμιστικά πλαίσια σε κάποιες περιπτώσεις για να είναι συμβατά με αυτές τις επιλογές. Ένα άλλο ζήτημα είναι η συντηρητική στάση και νοοτροπία απέναντι ε, σε, αυτή, σε αυτές τις επιλογές. Κυριαρχεί η νοοτροπία του πραγματικού κόστους, δηλαδή δικαιολόγηση και τεκμήρωση όλων των δαπανών άλλα πιο συγκεκριμένα σημεία που αφορούν καθέναν από τους τρεις βασικούς τύπους κόστους που προανέφερα. Σε κάποια κράτη-μέλη, για παράδειγμα, μας είπαν ότι τα κατόφλια, το ποσοστό πρέπει να εφαρμόζεται ε, στο κόστος για την ε, άμεσο, για, άμεσο κόστος για την επιστροφή έμεσων δαπανών είναι πολύ χαμηλό, δεν έχουμε ιστορικά δεδομένα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές λόγω των διαφορετικών παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και ε, εκεί ε, είναι το πρόβλημα με, τις μοναδιές, ε, με το μοναδιαίο κόστος και στα καταποκοπήν ποσά. Τι γίνεται αν η δραστηριότητα για την οποία ζητείτε επιστροφή με βάση ένα καταποκοπήν ποσό δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στη φάση του 80%, χάνεται όλο το ποσό, τι γίνεται λοιπά. Νομίζω ότι όλα αυτά εξηγούν γιατί ε, ιδίως τουλάχιστον οι δύο τελευταίοι τύποι δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί, αλλά ε, μόνο δειλά θα έλεγα ακόμη. Αυτά είχα να πω. Συνολικά νομίζω ότι είναι θετική εικόνα. Είναι θετική, πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, ό,τι αφορά την ε, δομήν καθοδήγηση, αλλά σίγουρα υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτιώσεων. Δύο πράγματα πρέπει. Πρώτον, να εμβαθύνουμε και να δούμε τι ε, τρει μεμονωμένε αυτέ τι επιλογέ απλοποιημένου κόστου. Μήπω χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, κάποιε τυποποιημένε επιλογέ ε, έτοιμε για τα κράτη-μέλη ή ε, κάτι που μας εξέπληξε σε πολλές από τις συνεντεύξεις και χωρίς να θέσουμε το ερώτημα μας είπαν Ιδίως σε σχέση με την εναρμόνιση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού, Κοινωνικού συγγνώμη, Ταμείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνω μας εξέπληξε ε, σε ό,τι αφορά τα πολυταμιακά ψηφιακά προγράμματα για την ε, ανάγκη απλούστευσης. Δηλαδή να έλθουν πιο κοντά τα δύο διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη το έργο μας. Συνεχίζεται. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μιχαήλοβα μου ζήτησε να διευθύνω λίγο τη συζήτηση καθώς έχει μια άλλη υποχρέωση. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Μπλόμαερ για την εισαγωγή σας για τις απλοποιημένες επιλογές ε, κόστους και η έκκλησή σας ε, για το πλαίσιο εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων που θα πρέπει να προσαρμοστεί παραδείγματος χάρη σε όσα αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Περιφερειακό Ταμείο είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα θέλαμε αλλά κάπου στη διαδρομή κολλήσαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κυρία Τετλινγκ της ε, Matrix και MBH για την ηλεκτρονική συνοχή και σε ποιο βαθμό μπορεί να μας ε, βοηθήσει. Κυρία Τέτλινγκ Σενχόφερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που αλλάξατε και τις ε, διαφάνειες. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τα πρώτα αυρήματα της μελέτης για την e-cohesion ηλεκτρονική συνοχή. Μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω εντάχει ποια είναι η λογική, τι σημαίνει αυτό το, αυτός ο όρος, τι ξέρουμε για την κατάσταση και να σας παρουσιάσω ορισμένα συμπεράσματα. Η πηγή, η βασική πηγή πληροφοριών είναι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και κάποια ερευνητική δράση δευτερογενής που έγινε με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς πάει η υλοποίηση. Ποιο είναι, ποια είναι η λογική, η έννοια της ηλεκτρονικής συνοχής. Ξεκινήσαμε με το δεδομένο ότι το διοικητικό κόστος είναι, θεωρούνται ότι είναι υπερβολικά υψηλά, ιδίω ό,τι αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση των έργων. Η, το e λοιπόν έχει σαν στόχο να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των δικαιούχων. Ένα από τα δέκα σημεία των ε, μεταρρυθμίσεων της ε, πολιτικής συνοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ως ορισμός είναι ότι η ηλεκτρονική συνοχή είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός των δικαιούχων και των διαχειριστικών αρχών αφενός και των διαχειριστικών αρχών άλλων προγραμμάτων που εφαρμόζουν ε, δραστηριότητες διαχείρισης και με τον ελεκτικό μηχανισμό. Έχει κοινούς κανόνες για την απλοποίηση της λογοδοσίας και πιο σωστής ε, λογοδοσίας των ταμείων. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να παρακολουθήσουμε πώς γίνεται η ηλεκτρονική συνοχή. Πρώτα απ' όλα ένα κράτος μέλος πρέπει να καταγράψει στην Συμφωνία Εταιρική Σχέση και στο πρόγραμμα δράση ΠΟΚ βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για τη μείωση της, ε, του διοικητικού βάρου, το πώ προτίθενται να υλοποιήσουν το σύστημα ηλεκτρονική συνοχή. Σε τακτή βάση γίνεται εξέταση της κατάστασης με την παρακολούθηση και υπάρχουν υγιές ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει θέση για την ηλεκτρονική συνοχή και τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις πρόοδου για την ηλεκτρονική συνοχή. Οι απαιτήσει της ηλεκτρονικής συνοχής έχουν, ε, αφορούν εκείνους που έχουν υπογράψει μια σύμβαση χρηματοδότηση, όχι τους ετούντες. Βεβαίως, τα κράτη-μέλη μπορεί να επεκτείνουν ωστόσο το σύστημα αυτό και στις αιτήσει για έργα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι ο κανονισμός κοινών διατάξεων και ο οδηγός δεν, πρέπει να, ζητούν τεχνικές απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι λογικό, διότι η ηλεκτρονική συνοχή δεν ήρθε εκ του ουρανού. Ε, υπήρξαν συστήματα που απλώς εξελίχθηκαν. Τα επιχειρησιακά περιφερειακά προγράμματα των κρατών μελών κατά συνέπεια μπορούν να επιλέξουν τον καλύτερο τρόπο για την πλήρη ανάπτυξη της έννοιας αυτής. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες ελάχιστες απαιτήσει. Μία από τις πιο σημαντικές είναι ένας κωδικός αναφορά. Μια, μια, φορά, μια φορά. Δηλαδή κάθε δικαιούχος πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του μία φορά και όχι περισσότερο. Υπάρχει και η έννοια της διαλειτουργικότητας. Δηλαδή σε ένα πρόγραμμα ένας δικαιούχος πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες αυτές άπαξ και τα θεσμικά όργανα πρέπει να αλλάζουν μεταξύ τους τις ε, πληροφορίες. Επίσης, ε, το ελεκτικό ηλεκτρονικό μονοπάτι πρέπει να, είναι, να συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα. Υπάρχουν και άλλες απαιτήσει για την αυθεντικότητα και επιστοποίηση των δεδομένων ε, και το πώς αποθηκεύονται τα στοιχεία. Πώς έχει κατάσταση τώρα το δεύτερο τμήμα. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες που έχουμε στη φάση αυτή για την κατάσταση. Η Συμφωνία εταιρική σχέση πρέπει να παράσχει λεπτομεριακή ενημέρωση για το πώς ε, προγραμματίζονται και εφαρμόζονται τα συστήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Τα, τα μισά από τα κράτη-μέλη έχουν δώσει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτό, τα άλλα μισά πολύ λιγότερο λεπτομεριακές ε, περιγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εικόνα για την ποιότητα του έργου και δεν μπορούμε να κλείσουμε αν η βασική πρόθεση για μείωση του διοικητικού βάρους των δικαιούχων υλοποιήθηκε ή όχι. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες συστημάτων. Κράτη-μέλη που έχουν ένα σύστημα αναταμείο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες συστημάτων ηλεκτρονικής συνοχής ανάλογα με το ταμείο που ισχύει. Άλλα κράτη-μέλη έχουν ένα σύστημα αναπεριφερειακή διοικητική μονάδα που επίσης πληρεί τις τα προπετούμενα για την ηλεκτρονική συνοχή αλλά ε, βρίσκεται καθοδόν, όχι στο τέλος. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ένα σύστημα για όλα τα ταμεία συνοχής και υπάρχουν και μια σειρά μεικτών συστημάτων όπου τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να ενσωματώσουν το Περιφερειακό, το Ταμείο, Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο, όλα τα υπόλοιπα είναι απ' έξω. Η έκθεσή μας θα σας παρουσιάσει τα προφίλ των κρατών μελών, λέγοντας ε, τι συστήματα υπάρχουν και κάποιες ε, περιλήψεις του πώς λειτουργούν. Αλλά εδώ βλέπετε έναν αριθμό κρατών με ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα στην αριστερή στήλη, ενώ στη δεξιά στήλη βλέπετε κράτη που έχουν μεικτά ή πολλά συστήματα. Τι μπορούμε να πούμε για την κατάσταση τώρα. Υπάρχουν τα συστήματα παντού, όπως ζητήθηκε να γίνει από τα κράτη-μέλη. Αλλά μεταξύ, φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, θεωρητικά εφαρμόζω και ουσιαστικά εφαρμόζω. Έχουμε κάποιες τέτοιες εμπειρίες. Στην πράξη η πρόκληση συνίσταται στην προσαρμογή που χρειάζεται για να ανεβάσουμε την, για να ανεβάσουμε τις αιτήσεις εκθέσεις εφαρμογής του 2016. Στη φάση αυτή γνωρίζουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη έδειξαν ότι είναι φιλόδοξα. Θέλουν να πάνε στις απαιτήσει που όπως είπα είναι αρκετά απλές. Κάποια κράτη εισήγαγαν περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα δικτών που ξεπερνούν το κοινό, τις κοινέ απαιτήσει. Αυτό διευκολύνει την αξιολόγηση. Υπάρχει ελπίδα προφανώς ότι η ηλεκτρονική συνοχή θα μειώσει το διοικητικό φόρτο. Υπάρχουν αξιολογήσεις που λένε ότι θα υπάρξει μείωση από 11% σύμφωνα με κάποιες μελέτες, άλλες ε, μελέτες είναι λιγότερο αισιόδοξες και μιλούν για μείωση 4 με 5%. Θεωρητικά είναι όλα αυτά ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε τι πραγματικό κέρδος υπάρχει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά είναι προσαρμοσμένα τα συστήματα και χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες. Σε ένα, σύστημα αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες που έχεις εφαρμόσει. Το ecohesion λοιπόν είναι εργαλείο. Αν δεν μειώσεις ωστόσο το διοικητικό φόρο στις διαδικασίες που ακολουθούνται δεν μπορεί να απλοποιήσεις ε, με την ηλεκτρονική συνοχή απλά και μόνο. Ένα εργαλείο είναι δηλαδή το e-cohesion. Κάποια μελη χρησιμοποιούν καινοτόμους τρόπους για να αναπτύξουν πλήρες ε, ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων. Κάποια άλλα κρατημέλη έχουν επεκτείνει το σύστημα και στις αιτήσει. Ένα σημαντικό βήμα για να διευκολύνουμε τη διοικητική, το διοικητικό βάρος. Βέβαια, το να υπάρχει απλώς ένα σύστημα δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να επιτύχουμε. Το να προχωρήσουμε σταδιακά σε μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση είναι προς όφελος της υφιστάμενης διαδικασίας. Το ερώτημα συμβάλλει στην απλοποίηση. Είναι δύσκολη η ερώτηση γιατί τα συστήματα η Cohesion έχουν σαν στόχο να, μειώσουν την επικάλυψη και, την, ε, και τον πολλαπλασιασμό των ε, τιμάτων για ίδια έγγραφα. Αν έχει ένα σύστημα, καταρχά θα υπάρξει μια αύξηση της, ε, του διοικητικού βάρους γιατί για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση του προσωπικού στο ξεκίνημα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους πριν αρχίσουμε να δρέπουμε τα θετικά αποτελέσματα. Ένα εμπόδιο που πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η εθνική νομοθεσία απαιτεί για παράδειγμα να υπάρχουν έντυπα ενώ η ηλεκτρονική συνοχή ως δεδομένο θεωρεί ότι δεν έχεις έντυπα σε χαρτί δηλαδή Αν λοιπόν υπάρχει έτοιμη, απέτηση για να υπάρχουν έντυπα κείμενα, δημιουργείται ένα θέμα. Επίσης θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει συνέχεια, να, να μην δίδεται συνέχεια στην ε, με, μόνιμη μελέτη της ανάγκης για μείωση του διοικητικού βάρους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τέτλινγκ Σενχόφα, ένα μικρό σχόλιο από μένα. Οπωσδήποτε οι προσδοκίες που είχαμε από την ε, ηλεκτρονική συνοχή, το e-cohesion, φαίνεται ότι στο θέμα της εφαρμογής και της κοινή διαχείρισης με τα κράτη-μέλη κάπου να κολλάνε. Και από την άλλη, επειδή κάθε κράτος θέλει να εφεύρει ξανά τον τροχό από μόνο του και δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εμείς θέμε να υπάρχει μια συγκρισιμότητα της εφαρμογής των ε, προγραμμάτων, αλλά αυτό δεν γίνεται εκτός εάν τα κράτη-μέλη μας ε, δίνουν τα δεδομένα τους με τρόπο συγκρίσιμο. Είμαι και στην Επιτροπή Ενέχου του Προπολογισμού και πραγματικά μας λυπεί αυτό. Αλλά εκφράσατε και μόνοι σας ε, την ελπίδα να ε, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και να έχουμε κάποιες βελτιώσεις ε, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τώρα ο καθηγητής Τζον Μπάχτλερ έχει τον λόγο. με ένα θέμα το οποίο φαίνεται κάπως ως όνειρο θερινής νυχτός δεδομένων των πάρα πολλών κανονισμών και ελεγκτικών μηχανισμών που υπάρχουν. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως λέτε, ο τίτλος είναι κάπως προκλητικός, δηλαδή αν η απλοποίηση είναι απλά μόνο στη φαντασία μας. Θα ήθελα λοιπόν κάπως να διευρύνω την οπτική μας γωνία όσον αφορά τα ζητήματα της αυλοποίησης. Θα ήθελα κατά βάση να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα, σε δύο είδη ζητημάτων. Το ένα είναι τι πρόοδο έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής στην τρέχουσα περίοδο μετά τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και δεύτερον πού πρέπει να πάμε στο μέλλον. Ποιες θα είναι οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, βασίζομαι σε μια έρευνα των διαχειριστικών αρχών που έγινε σε 15 κράτη-μέλη υπό την αιγίδα του δικτύου QNET, ε, στο οποίο ανήκουν 18 διαχειριστικές αρχές από τις 15 αυτές χώρες. Είναι ένα δίκτυο το οποίο υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και εστιάζει σε πρακτική ανταλλαγή πληροφοριών και η παρουσίασή μου αντλεί στοιχεία από μια συζήτηση και έρευνα δηλαδή που είχε αναφερθεί και στην τελευταία τους ε, συνεδρίαση και υπάρχει μια ενημέρωση στα έγγραφά σας. By Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας τι πρόοδο έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα και οι δύο παρατηρήσεις που μόλις έγιναν τώρα έτσι θα τεθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναλυφθεί για την απλοποίηση και νομίζω πως το πρώτο το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε όπως έκαναν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος υπό την έννοια ότι οι μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς Θεωρείται ότι έχουν βελτιώσει την ε, εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων. Βλέπετε εδώ πέρα την άποψη των διαφόρων διαχειριστικών αρχών για το εάν συμφωνούν ε, με το ότι όλα αυτά τα μέτρα, τα καταποκοπήν ποσά, η ηλεκτρονική διαχείριση κτλ. Ε, έχουν κάνει κάποια διαφορά. Στα αριστερά λοιπόν βλέπετε αυτά τα οποία θεωρείται ότι έχουν ε, συνεισφέρει περισσότερο. Ειδικά τα το απλοποιημένο κόστος, τα καταποκοπήν ποσά, οι μικτές ε, ε, διαχειριστικές διατάξεις, οι κοινέ διαχειριστικές διατάξεις θεωρούνται πιο χρήσιμα μέτρα. Στην άλλη άκρη του φάσματος υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη για το πόσο συνεισφέρουν στην απλοποίηση μέτρα όπως η τοπική ανάπτυξη και τα σχέδια δράσεις. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα και βλέπουμε πως κάποια κράτη-μέλη δεν υιοθετούν τις διατάξεις αυτές πέρα από το απολύτως απαραίτητο. Βεβαίως αναγνωρίζουμε πως τα μέτρα αυτά είναι νέα και ίσως ακριβώς να είναι επιφυλακτικοί γιατί δεν τα γνωρίζουν. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών ως αντίδραση στις ε, νέες διατάξεις. Βλέπουμε σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά την απλοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας και την εναρμόνιση των κανόνων ε, και των ε, εντύπων των αιτήσεων σε πολλά κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τους ε, μηχανισμούς εκτέλεσης ε, π.χ. ένα ενιαίο site, ε, τυποποιημένες αιτήσει και διαδικασίες και περισσότερη στήριξη στους δικαιούχους για να μπορούν να δουν τι γίνεται με την αίτηση. Υπάρχει σημαντικός βαθμός απλοποίησης της αρχιτεκτονικής του προγράμματος και μία μείωση ε, στον αριθμό των προγραμμάτων ε, και των ε, εφαρμοστικών φορέων. Και τέλος βλέπουμε πως υπάρχει μία απλοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης. Όμως, αν τα δούμε λίγο από απόσταση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η απλοποίηση, η το περιθώριο για απλοποίηση πρέπει να το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο των διαδοχικών ε, ρυθμιστικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα σε διαδοχικές μεταρρυθμίσεις μετά την μεταρρύθμιση των ε, διαρθρωτικών ταμείων το 1988 και αυτή η διαφάνεια μας δείχνει τα διάφορα στρώματα θα έλεγα διατάξεων που έχουν εισαχθεί στις διάφορες ε, μεταρρυθμίσεις και βεβαίως κάθε φορά είχαμε και περισσότερη πολυπλοκότητα. Παραδείγματο χάρη, ενώ υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να υπάρχει μια στρατηγική συνοχή, μια θεματική συγκέντρωση για να επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα, το κάθε ένα από αυτά φέρνει έχει ταυτόχρονα και νέε προκλήσεις, π.χ. συνεργασία με νέους δικαιούχους ε, ή όσον αφορά την στρατηγική συνοχή το ότι απαιτείται, απαιτούνται νέες θεσμικές σχέσεις. Τώρα, για να περάσουμε από την θετική προόδο στα ζητήματα τα οποία ανησυχούν τις ε, διαχειριστικές αρχές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους ε, τίτλους. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αυτά τα οποία θα λέγαμε διαρθρωτικά και συστημικά ζητήματα και πρώτο πρώτο σε αυτά είναι η περιπλοκότητα των διαδικασιών καθορισμού των ε, διαχειριστικών αρχών και των αρχών οι οποίες πιστοποιούν και αυτό βεβαίως ήταν μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία και βεβαίως εμποδίζεται έτσι η πρόοδος ε, όσον αφορά την εφαρμογή. Όσον αφορά λοιπόν τις ε, διαχειριστικές αρχές, κατά την άποψή τους, τους δυσκολεύει και η μη εναρμόνιση των κανόνων και η αντίληψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο εν μέρη στα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και στους ε, Τομεί της πολιτικής ε, συνοχής και στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Και υπάρχει κάποια ανησυχία για τις επιπλέον απαιτήσει που έχουν εισαχθεί ειδικά με τις νέες πρωτοβουλίες που ανέφερα. Κάποιες άλλες ανησυχίες ε, των κρατών μελών αφορούν ε, την ερμηνεία που δίδεται και την καθοδήγηση. Και εδώ πέρα η βασικότερη ενισχύα είναι η έλλειψη νομικής βεβαιότητας που σχετίζεται με διάφορους παράγοντες αλλά ειδικά με το ότι είναι πάρα πολλά τα κείμενα ή κανονισμοί και το ότι υπάρχει μια ασυνέπεια μεταξύ αυτών των κειμένων. Όταν μιλάμε δε για την νομική ασφάλεια που και που αναφέρεται επίσης ο υπερθεματισμός των κρατών μελών τα οποία συχνά κατηγορούνται ότι προσθέτουν δικά τους πράγματα πάνω στους κανονισμούς. Δηλαδή βάζουν τα κράτη-μέλη διατάξεις ε, με στόχο να προστατεύσουν τα προγράμματα από τον δημοσιονομικό έλεγχο και για να υπάρχει κάποια νομική βεβαιότητα. Υπάρχει επίσης ανησυχία για το καθεστώς ε, των κατευθυντήριων γραμμών της Κομισιόν, οι οποίες βεβαίως είναι καλοδεχούμενες, αλλά τι είναι αυτά, είναι συμβουλές, είναι πρακτικέ πρακτικές, είναι ιονοί κανονισμοί που τελικά θα τα βρουν μπροστά τους οι διαχειριστικές αρχές τη στιγμή του ελεγχού, όπως είπε και ο κύριος Μπλομάιερ, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τις επιλογές του απλοποιημένου κόστους και των ποσών κατά Ένα άλλο θέμα αφορά τις διαδικασίες ελέγχου και εδώ πέρα περνάμε σε κάποιες προτάσεις για αλλαγή και δεν κοιτάμε μόνο τα προβλήματα αλλά και το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις. Και υπό τον τίτλο των ελεγκτικών διαδικασιών Μία από τις ε, προτάσεις που έκανε μια διαχειριστική αρχή είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύμφωνο κοινή ερμηνεία μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελεγκτικών αρχών για να υπάρχει κάποια νομική βεβαιότητα για να μειωθούν οι προκλήσεις ε, που υπάρχουν όσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην παραγωγή. Επίσης υπάρχει το αίτημα να υπάρχει περισσότερη αναλογικότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Αναλογικότητα η οποία θα βασίζεται στο μέγεθος της χρηματοδότησης, στο ύψος της χρηματοδότησης, στον κίνδυνο επέλευσης σφάλματος και στο ποσό βεβαίω, το οποίο διακυβεύεται. Και ερχόμαστε άρα στο τρίτο θέμα, την τρίτη πρόταση, δηλαδή ότι υπάρχει περιθώριο απλοποίηση των πολλαπλών επιπέδων ελέγχου, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν εθνικά συστήματα τα οποία λειτουργούν και όπου υπάρχει ένα ιστορικό το οποίο αποδεικνύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει λιγότερη ανάγκη ελέγχου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης για το μέλλον θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο εναρμόνισης των κανόνων και της ερμηνείας στο έγγραφο ενημέρωσης που σας δώσαμε και στην έκθεση που υπάρχει πίσω αυτό υπάρχουν κάποιες προτάσεις για κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν απλά και γρήγορα απλές αλλαγές ε, με μικρές ρυθμίσεις και ένα σημαντικό τομέα για να αναζητήσουμε αλλαγές, ειδικά για μετά το 2020, είναι το που υπάρχει περιθώριο ευθυγράμμισης των ε, ρυθμιστικών απαιτήσεων διάφορων πολιτικών. Και ένας τομέα ε, είναι αυτός ο οποίο ανισχύει περισσότερο τι διαχειριστικέ αρχές. Είναι η σχέση της πολιτικής συνοχή με την πολιτική ανταγωνισμού. Παραδείγματο χάρη, αν η έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετίζεται με διαδικασίες κοινοποίησης στην Κομισιόν. Και τέλος, για να διευρύνουμε λίγο κάπως την οπτική μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς όσον αφορά τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν εντός του υφιστάμενου συστήματος κοινή διαχείρισης, γιατί υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να γίνει με την υφιστάμενη διαχειριστική δομή. Βεβαίω η κοινή διαχείριση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ε, δεν λειτουργεί όσο αποτελεσματικά θα θέλαμε. Και ειδικά καθώς τώρα είμαστε στην περίοδο του να σκεφτόμαστε το τι θα γίνει στο μέλλον μετά το 2020, νομίζω πως μια σημαντική σύσταση είναι να χρησιμοποιήσουμε τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τους ε, κοινούς ε, ευρωπαϊκούς κανόνες εκεί όπου χρειάζονται και να υπάρχει περισσότερη ευελιξία για τα εθνικά συστήματα και κανόνες ε, όπου υπάρχει βεβαίως διασφάλιση από τον κίνδυνο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και υπάρχουν και περαιτέρω πληροφορίες βεβαίως για αυτά τα οποία ανέφερα. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για αυτά τα οποία μας είπατε και για το ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο στην φαντασία μας η απλοποίηση αλλά για το ότι υπάρχουν προτάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της κοινής διαχείρισης ως μια ε, δυνατότητα απλοποίησης και σας ευχαριστώ. Οπότε, αφού ακούσαμε τους ειδικού, περνάμε στην σκοπιά αυτών που ασχολούνται με την εφαρμογή τα κράτη-μέλη δηλαδή και τις περιφέρειες. Ξεκινάμε με την κυρία Σαντάλ Μωρό η οποία είναι αρμόδια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα την περιφέρεια Όβερν, Ροδανού και Αλπέων. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε και ως ε, διαχειριστική αρχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε καθημερινές επαφές ε, με τους ε, εκτελούντες έργα και θέλουμε να κατανοήσουμε και να δούμε πώς εφαρμόζονται οι εθνικοί, περιφερικοί και ευρωπαϊκοί κανόνες. Ε, στην Οβέρνη Ροδανό Άλπης ε, είμαστε υπεύθυνοι για πολλά επιχειρησιακά προγράμματα ένα για τη συνεργασία και τρία για την περιφερειακή πολιτική, πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ διαθωτικά κονδύλια για την περιφέρεια αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είμαστε προσιλωμένοι, αλλά και πόσο πρέπει να προσέξουμε την εφαρμογή των κανόνων. Όπως γνωρίζετε στη Γαλλία Πρόσφατα είχαμε δύο πολύ σημαντικές αλλαγές. Αφενός ε, τα περιφερειακά συμβόλαια, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε διαχειριστική αρχή ε, για την περίοδο 14-20 ε, μετά από μια μακρά περίοδο που την ευθύνη αυτή την είχε το κράτος. Οι περιφέρειες δεν είναι ότι δεν είχαν εμπειρία γιατί ήταν ενδιάμεση στις δύο προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Η ευθύνη όμως της διαχειριστικής αρχής, η διαρχή του ελέγχου είναι στην τοπική αυτοδίκηση το 2014. Το 2015 είχαμε την ε, εδαφική μεταρρύθμιση στη Γαλλία μειώθηκαν ε, κατά το ίμιση οι περιφέρειες και από τον Ιανουάριο εμείς είμαστε πλέον μία περιφέρεια, η Ροδανός, Άλπης και η Οβέρνη. Για μας αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να διερωτηθούμε και για το ποιος είναι ο ρόλος της διαχειριστικής αρχής ιδίως σε ό,τι αφορά τους κυρίους έργου διότι όπως βλέπετε εδώ και όπως υπόθηκε και προηγουμένως η διχειριστική αρχή ουσιαστικά είναι ένα γρανάζι, ένας ε, κρίκος της αλυσίδας, ασκεί έλεγχο ε, ε, σε ό,τι αφορά τους ε, εργολάβους, αλλά ε, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αλυσίδα του ελέγχου υπάρχει και ο εργολάβος ε, και νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε στο επίκεντρό μας την απλούστευση της διαχείρισης των κονδυλίων των διαρθωτικών ταμείων. Το θέμα που πρέπει να σας ε, παρουσιάσω σήμερα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το διοικητικό ε, βάρος υπέρ των δικαιούχων. Είναι δύσκολο να σας πω συγκεκριμένα τι κάνουμε, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, αλλά ε, μπορώ να σας πω και κάποια σχόλια σε σχέση με ό,τι άκουσα, παραδείγματος χάρη για το e-cohesion και κυρίως ε, την αϊλοποίηση των διαδικασιών, ε, δηλαδή για την εξοικονόμηση ε, και σε πόρους αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε ό,τι αφορά ε, τον εργολάβο, ε, θέλουμε να είναι απέναντι μας για να μας εξηγήσει ποια είναι τα προγράμματα του, ποιοι είναι οι στόχοι του ε, και πώς θέλει να τους επιτύχει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη η μέθοδο υλοποίησης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για αυτή την περίοδο είχαμε έναν εργολάβο, έναν ανάδοχο για ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό σχέδιο για κάποια σταθμομέτρηση και στο πέστο του επιχειρησιακού προγράμματος στείλαμε την σύμβαση. Ο ανάδοχος διάβασε τη σύμβαση, είδε ότι ένα άρθρο ε, του ζητούσε ρητός να διατηρεί ε, σταθμούς ε, την επένδυσή του δηλαδή για πέντε χρόνια μας πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κοιτάξτε είναι πειραματική η δική μου σταθμή τους κρατώ για δύο χρόνια και μετά δεν ξέρω τι θα τους κάνω διότι είτε ε, Πρέπει να ξέρω τι θα γίνει με το σχέδιο. Θα αποτύχει, θα πετύχει. Δεν μπορώ να σα πω από τώρα αν θα κρατήσω ή δεν θα κρατήσω αυτού του ε, σταθμού. Και έτσι επαναπρογραμματίστηκε το σχέδιο και τελικά χρηματοδοτήθηκε ε, με το, από τον προπολογισμό του πλησιακού προγράμματο. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, πρέπει να αγωνιστούμε κατά της κατάσταση ε, των επιχειρήσεων και των δράσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι όμως κατάλληλο για ε, project ε, στον τομέα της καινοτομίας ή πειραματισμού, όταν αντιλαμβάνεται ρίσκο δηλαδή από τον υπεύθυνο για την εκτέλεση ενός έργου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τον ανάδοχο των δυνητικών να τον συναντήσουμε και να δούμε τι ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιο είναι ο τρόπος εφαρμογής του ε, project. Επίσης, όταν μιλάμε για απλούστευση, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τις κρατικές ενισχύσεις. Το θέμα μας ανησυχεί ιδιαίτερα και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, ήδη ακούσατε τις επιλογές για το απλουστευμένο κόστος. Είναι μια σημαντική πρόοδος για εμάς. Το επικροτούσαμε γιατί να κάτω το περιμέναμε. Η συμβατότητα της εφαρμογής ορισμένων ε, μηχανισμών κρατικών ενισχύσεων με το απλουστευμένο κόστος δεν έχει παληθευτεί ότι ισχύει. Και επειδή θέλουμε ο ανάδοχος να μην μας δίνει πια όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουμε αυτές τις αποστευμένες επιλογές, όμως όταν μιλάμε για προγράμματα που έχουν να κάνουν με την καινοτομία, με την οικονομία, ο κανόνας ε, που εφαρμόζεται ε, συνεπάγεται ρίσκο, κυρίως για τον ανάδοχο. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, όχι. Εμείς προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε την αρχή της εμπιστοσύνης προς τον δικαιούχο. Υπάρχουν κάποια ερευνητικά κέντρα, κάποιες ΜΜΕ που καινοτομούν ιδιαίτερα και που μπορούν να υποβάλουν για την ίδια περίοδο προγραμματισμού περισσότερα από το Όταν κάνουμε την επιλογή στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματο, επιλέγουμε ε, μία επιχείρηση, ένα project δηλαδή, ανάναδοχο και αν διαπιστώσουμε ότι εκεί δεν έχουμε πρόβλημα και ότι εφαρμόζεται σωστά, τότε αποφασίζουμε να μην ελέγξουμε την επόμενη χρονιά τον εργολάβο για οποιαδήποτε άλλη είδους ε, επιχείρηση που είναι εκτός του σχέδιου ελέγχου. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες ελέγχου, αλλά εμείς ως διαχειριστική αρχή προσπαθούμε να ελαφρύνουμε αν θέλετε το βάρος των ελέγχων. Και να πω κάτι ακόμη για τους ελέγχους γιατί έχουμε εμπειρία που σχετίζεται με την ευθύνη μας ως ε, διαμεσολαβητή, ως ενδιάμεση φορέα στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Λυπούμε γιατί δεν γίνεται διάκριση μεταξύ απάτης και σφάλματος. Όταν έχουμε μια οργάνωση, ε, ένα, μια μικρή επιχείρηση, μια τοπική αρχή, αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν αυτό τον κικαιώνα ε, κανονισμό που και εμείς σχολευόμαστε, να καταλάβουμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα μπορούν να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Ε, μικρή επιχείρηση μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος γιατί μπορεί να μην τήρησε την προθεσμία, μπορεί να ήταν ο αριθμό των ημερών μικρότερος από τον νομικό υποχρεωτικό αριθμό κτλ. Και άλλο ότι ήθελε σκοπίμως ε, να ε, πάρει κάποια κονδύλια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ναι, ένας εργολάβος έχει και το δικαίωμα στο σφάλμα. Μπορεί να κάνει λάθος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τιμωρηθεί ε, και να του επιβληθεί οικονομικό πρόστιμο αν χάνει τα επιδιακόμενα αποτελέσματα. Και επίση έχουμε αναστρέψει το βάρο τη απόδειξη. Δηλαδή, όταν εμεί ελεγχόμαστε τελικά, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν διαπράξαμε σφάλματα. Ο ελεγκτή δηλαδή έρχεται και μα λέει, μάλλον έχετε κάνει ένα σφάλμα και θα το βρω. Το ίδιο κάνει και στον ε, ανάδοχο, στον εργολάβο. Όμω ο εργολάβο, ε, ένα ε, επικεφαλή μια μικρή επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση, τι θέλει. Θέλει απλά να γίνει μια παρέμβαση για να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο που έχει αναλάβει. Τελεία και πάλι. Αν θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε σε ένα ε, συνεκτικό ποσοστό σφάλματος σε σχέση με αυτά που βλέπουμε επιτόπου, θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ σφαλμάτων και απατών. Έχουμε περιθώριο σφάλματος, μάλλον ποσοστό σφάλματος 2% και αν ε, έχουμε αυτό το 2% το τιμωρεί η Κομισιόν. Είναι πολύ δύσκολο, δύνατον με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία να μείνουμε σε αυτό το 2%, το συντελεστή σφάλμα το 2%. Ε, μηχανικά δηλαδή, οι διαχειριστικές αρχές δέχονται να μην λάβουν το σύνολο του προϋπολογισμού, διότι ένα μέρος θα διορθωθεί ε, κατά αποκοπή. Επομένως, αυτά είχα να πω. Δεν μπορώ να σας ε, πω περισσότερα, γιατί είπε πολύ διεξοδικά ο συνάδελφος για τις επιλογές, ε, τις στευμένες επιλογές κόστους. Πράγματι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αποσταυμένου κόστους και έχουμε κάποιες, κάποιους προσανατολισμούς. Καθοδήγηση. Έχουμε ένα άρθρο του κανονισμού, 24 σελίδες, ε, η καθοδήγηση έπειτα επεξηγήσεις. Γιατί ένα απλό άρθρο να χρειάζεται 24 ε, σελίδες επεξήγησης. Τέλος, εν κατακλείδη, νομίζω ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ε, που δεν την έχουν πια τα κράτη-μέλη ή ε, οι τοπικές αρχές. Εμείς έχουμε το γενικό, ε, το γενικό καταστατικό μας ε, που μας υποχρεώνει να ακολουθούμε κανόνες και έχουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους εθνικούς, από τη στιγμή που ζητούμε πεκά κονδύλια γιατί να ελεγχόμαστε περισσότερο όταν, από όταν ζητούμε κρατικά κονδύλια από το κράτος στην περιφέρεια ή από κάποιο άλλο φορέα. Επίσης, η αρχή της επικουρικότητας που εφαρμόζεται γενικά στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής εφόσον εκχωρεί η Κομισιόν στα κράτη-μέλη που και αυτά μπορούν να εκχωρήσουν αρμοδιότητες σε άλλες ε, ε κάτω του εθνικού επίπεδου ε, αρχές θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας ότι αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδύλων. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Frau Moreau. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα στην περιφέρεια αναφερθήκατε σε ένα ευαίσθητο ζήτημα που μας απασχολεί δηλαδή τι είναι το σφάλμα είπατε ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και πρέπει να δούμε πού είναι τα λάθη και πού αρχίζουν οι απάτες και πώς τα αντιμετωπίζουμε και οπωσδήποτε οι ελεγκτικές ε, διατάξεις είναι διαφορετικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό βεβαίως ξανά δυσκολεύει την δουλειά των αρχών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αφού λοιπόν ακούσαμε την κυρία Μωρό από το δυτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα θα ακούσουμε τον Υφυπουργό του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, της Πολωνίας, ε, τον κύριο Πάβελ Οράνζ. Πρόσον πάντα. Φίλεν τάγκ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάσω την εμπειρία μου. Ήμουν υπεύθυνο ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Πολωνία από τότε που εντάχθηκε η Πολωνία στην Ένωση. Η παρουσίασή μου λοιπόν εν βασίζεται στην εμπειρία μου ως ε, υπαλλήλων στην διοίκηση. Να σας δώσω καταρχάς κάποιες λεπτομέρειες ή την γενική προσέγγιση που υιοθετήσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κατόπιν θα μιλήσω για τα βήματα προς τα μπρος, τα βήματα προς τα πίσω και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης. Όταν διαπραγματευόμασταν ε, τις νέες ε, χρηματονομικές προοπτικές υπήρχαν δύο μορφές αφήγησης. Ένα, να απλοποιήσουμε. Δύο, ένας προσανατολισμός προς το αποτέλεσμα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στις δύο αυτούς τομείς που έπρεπε να αντιμετωπιστούν στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν βλέπουμε τις διαπραγματεύσεις και την έκβασή τους μπορούμε να πούμε ότι κάποιος σπόρος εσπάρει. Αλλά όταν σπείρεις τον σπόρο, τι βγάζεις, αυτό είναι το ερώτημα που έπρεπε να θέσουμε. Όταν βλέπουμε την κατάσταση και αξιολογούμε τις διαπραγματεύσεις ως Πολωνός εγώ δηλαδή, για πρώτη φορά θα μπορούσα να πω ότι εφαρμόστηκαν κάποιοι μηχανισμοί με έμφαση στο αποτέλεσμα. Κάποιοι από αυτούς όμως σε πολύ γενικό επίπεδο. Οι των προτέρων ε, προϋποθέσεις, το εξάντε conditionality που λέμε, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος παρέμβασης, δεν είχε γίνει ευπρόσδεκτη από μένα και τους συναδέλφους, αλλά δεν εφαρμόστηκε η πρόθεση των χρηματοοικονομικών ε, εργαλείων. Πιστεύουμε ότι είναι στομέα που δεν έτυχε πλήρους εκμετάλλευσης από τα διαθροντικά ταμεία και μπορεί να είναι ελκυστικός για τις διαχειριστικές αρχές. Η ευρύτερη εφαρμογή των SEOs και η υποχρεωτικότητα, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους ε, επίσης είναι κάτι χρήσιμο, η εισαγωγή κοινών προγραμμάτων δράσης που προσανατολίζονται προς τις επιδόσεις. Ε, μια αλλαγή δηλαδή της γενικής κουλτούρας που στην ουσία κάνει απλό έλεγχο των τιμολογίων αλλά που θα βλέπει τα αποτελέσματα. Είχαμε αλλάξει κάποια πράγματα, αυξήσαμε τα ανώτατα όρια, τα, τα κατώτατα όρια για κάποια έργα. Όλα αυτά είναι ένα βήμα προς τα μπρος που βοηθάει την, ε, ε, τα κέρδη. Εισάγαμε επίσης τους flat rates, τους, τους ενιαίους συντελεστές σε κάποιους τομείς. Επίσης χρησιμοποίησαμε αλγόριθμους. Μια τέτοια προσέγγιση δηλαδή που θεωρήθηκε πρόσδεκτη. Το ερώτημα βέβαια είναι οι υποσχέσεις ή κάποιες από αυτές σε τι βαθμό υλοποιήθηκαν. Αυτό που βλέπουμε είναι, ωραία, άλλαξε η αφήγηση, αλλά όχι τόσο η πρακτική. Όταν βλέπουμε τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, τις διαδικασίες που ακολουθούνται, δεν άλλαξε τίποτα στην πραγματικότητα. Λυπάμαι γιατί είμαι υπεύθυνο συντονιστή τώρα στην ε, Πολωνία, αλλά πραγματικά καταλαβαίνω πόσο στοιχίζει να υποβάλουμε, να επιβάλλω στους ε, υφισταμένους και συνεργάτες μου να ακολουθήσουν μια προσέγγιση SEO διότι είναι πάντα η τακτική ότι με το γνωστό πάμε καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα πούν τώρα οι ελεγκτές. Όλοι έχουν καταλάβει ότι είναι δύσκολο να, πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Επίσης, σε, κυρίως σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών, στα ενδιάμεσα σώματα. Οι καινοτόμες ιδέες ε, συγκρούονται με αυτά τα προβλήματα. Όταν έρχεται ο ελεγκτής δηλαδή, πώς το εξηγούμε ότι παρεκτράπημεν κατά κάποιο τρόπο από τα περιγεγραμμένα στον οδηγό. Αυτά τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τις ασυμβατότητες. Η πρωτοβουλία για το εισόδημα των νέων η... στην Πολωνία Έχουμε μια σειρά προγραμμάτων ε, εγγύηση νέων. Δεν, τα έξι από αυτά δεν είναι επιλέξιμα, αλλά εμεί είπαμε να δώσουμε έμφαση στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασία και τα υπαγάγαμε. Έχουμε λοιπόν οκτώ επιπρόσθετους δείκτες για τις 29 περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για την πρωτοβουλία νέων και 28 επιπρόσθετοι δείκτες δεν παρέχουν ε, προστιθέμενη αξία. Δεν έχουν δηλαδή νέα στοιχεία σε σχέση με, τα τυπικά, με τους τυπικούς δείκτες του κοινωνικού ταμείου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε μια εμπειρία ελέγχου από την Επιτροπή για το Youth Employment Initiative, την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Εμείς είμαστε στη διαδικασία συζήτησης για το θέμα αυτό με την Επιτροπή, αλλά Μία από τις βασικές συστάσεις προς την Πολωνία ήταν τα άτομα που είναι απαθή, αδύνα, που δεν μπορούν να καταχωρηθούν ως ε, ετούντες εργασίας στα γραφεία ευρέσεως εργασίας, να τους προσεγγίσουν μικιό για να τους, εάν είναι επιλέξιμοι, να είναι κάτω από τα 28 για παράδειγμα, και να ετοιμαστεί ένα κείμενο που να τεκμηριώνει ότι είναι άνεργοι. Όταν ρωτάμε λοιπόν γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι άτομα που μετέχουν στο σχέδιο περνούν χρόνο σε training ε, γιατί να Τέλο γιατί να χρειάζεται να αποδείξουν ότι είναι άνεργοι ή ότι δεν απασχολούνται. Γιατί άμα απασχολείσαι, προφανώ μπορεί να πα σε χρόνο, σε κατάρτιση ή σε, σε μια πρακτική. η ιδέα, μάλλον η, ο παραλογισμό αυτός... αλλάζει σε ψηλά επίπεδα, αλλά όσο κατεβαίνουμε στην ιεραρχία, οι, οι παραμένουν. Άλλο θέμα. Κανόνες κρατικών ενισχύσεων ε, και δραστηριότητε που παρέχουν εισόδημα, το revenue enhancing ε, ε, policies. Εκεί βλέπουμε ότι η πολιτική συνοχή είναι το πεδίο μάχης όλων των κανονισμών της Ένωσης. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να δούμε τι θα εφαρμόσουμε. Κανόνες τις πολιτικές συνοχής, κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, άλλους κανόνες που επιβάλλονται από άλλες αρχές ή ελεγκτικά όργανα. Ωραία λοιπόν η ιδέα της ηλεκτρονικής συνοχής. Μπράβο, μπράβο. Αλλά απλοποιούμε τις διαδικασίες και καθιστούμε τις διαδικασίες ή ηλεκτρονικές ή κάνουμε ηλεκτρονικές συμφιστάμενες διαδικασίες. Αυτό είναι το θέμα. Λέμε λοιπόν ότι πολύ ωραία η ηλεκτρονική συνοχή για τους δικαιούχους και τα λοιπά, αλλά άμα δείτε τον κανονισμό της Επιτροπής που είναι όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεφούν. ο κατάλογος είναι τεράστιος και τα περισσότερα στοιχεία πρέπει να τα δώσουν οι δικαιούχοι. Καλή ιδέα, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνονται πολλά. Τώρα, πώς θα βγούμε από αυτό το λαβύρινθο. Να αλλάξουμε φιλοσοφία. Φιλοσοφία υλοποίησης. Είπε κάποιος ήδη ότι πολλοί θεωρούν πως ε, το κόστος, το πραγματικά καταβληθέν κόστος, είναι πολύ καλό γιατί μπορεί να μην κερδίσουμε τίποτα αλλά παίρνουμε τα λεφτά μας. Το λένε αυτό πολύ. Εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να στραφούμε στα αποτελέσματα για να εντάξουμε τις διαδικασίες στην αυτή φιλοσοφία. Αλλιώς θα Βλέπουμε τη συμμόρφωση με τους δημόσιους τομείς, ε, διαφορετικούς, ε, διαφορετικά αποτελέσματα κλπ. Οι δημόσιες συμβάσεις, τα SEO, είναι οι κλασικά παραδείγματα. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διαδικασία όταν έχουμε μεγάλο κομμάτι κρατικών συμβάσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε τα αποτελέσματα, την παραγωγή, όχι την τήρηση των κανονισμών σαν βασικό μας στόχο. Το δεύτερο θέμα, um, uh, το οποίο νομίζω ταυτίζεται με πολλές από τις απόψεις που εκφράστηκαν, να μην ε, αθρίζουμε κανόνες μετά από κάθε έλεγχο. Γιατί αυτό που μας φοβίζει είναι ότι σε πέντε χρόνια θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι κανόνες που δεν θα προκύπτουν από κανονισμούς αλλά που θα επιβάλλονται σταδιακά από τους ελεγκτές. ο τελικός κριτής είναι πάντα ο ελεγκτή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν έχετε λοιπόν στην Επιτροπή κάποιον ο οποίο στην Επιτροπή Ελέγχου που μπορεί να παρέμβει μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των ε, ελεγκτών και να ε, τους πει κοιτάξτε την πραγματικότητα ρε παιδιά δείτε λίγο την κοινή λογική θα ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό η παράγωγη νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που το ανέφεραν άλλοι. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπρος που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε πλήρως. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες για το τι ποσοστό γίνεται CSCO. Αυτό που θέλω όμως ε, να δω είναι να, να λάβει ενεργό ρόλο επιτροπή. Υπάρχει το άρθρο 40 παράγραφος 1 στον κανονισμό του, του, του Κοινωνικού Ταμείου που επιτρέπει στην επιτροπή να υιοθετήσει πανευρωπαϊκές επιλογές μείωσης κόστους ε, με κανονισμούς. Αν δείτε λοιπόν το Κοινωνικό Ταμείο θα διαπιστώσετε ότι Έχουμε πολλές ε, μορφές ε, μείωσης ε, του κόστους. Στο Λεωνάρντο, στο Εράσμους υπάρχουν μορφές μείωσης του κόστους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... και στην πολιτική συνοχή. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθούν επιλογές μείωσης του κόστους. Το ίδιο θα πρέπει να προσθεθεί και στο ΦΕΝΤΕΡ, στο Περιφερειακό Ταμείο. Αυτό θα πει εναρμόνιση κανόνων όχι ομοιογενοποίηση. Δεν θα έπρεπε να ταυτίζουμε τους δύο όρους. Αυτή είναι η δική μας εμπειρία στην Πολωνία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εξαιρετική παρουσίαση. Και θα ξαναδώσω τώρα τον λόγο στην Πρόεδρο. Thank you very much. Thank you for the support, uh, Mr. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσέλερ και σας ευχαριστώ για την ε, για τις παρουσιάσεις. Λοιπόν, συνάδελφοι, δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν και της Επιτροπής των Περιφερειών ή να μαζέψουμε προτάσεις ε, από τους ε, συναδέλφους και μετά να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις. Θέλετε να θέσετε ερωτήσεις, σχόλια τώρα ή να ακούσουμε την Κομισιόν. Καλώς, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Περίμενα ερωτήσεις, οφείλω να πω. Προφανώς ε, αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα των θεμάτων αυτών. Κάπου κάποια στιγμή, κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες υπάρχει μια συνεδρίαση για την απλοποίηση. Μάλιστα η μονάδα μου μόλις άλλαξε το όνομά της σε καλύτερη εφαρμογή. Ίσως θα έπρεπε να γίνει η απλούστερη εφαρμογή. μια ακόμη καλύτερο. Πρέπει να πω πως κάθε φορά που έρχομαι σε αυτές τις ε, συζητήσεις αισθάνομαι την ανάγκη να υπεραμεινθώ των πρακτικών της Κομισιόν γιατί συχνά υπονοείται ότι όλες αυτές οι δυσκολίες και περιπλοκές οφείλονται στην Κομισιόν και εμεί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το βλέπουμε σε μια κοινή προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων και όλοι μαζί να προωθήσουμε την απλοποίηση. Να σας πω λίγο λοιπόν πώς τα βλέπει η Κομισιόν. Χωρίς να δραματοποιούμε την κατάσταση, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση πως ε, βρισκόμαστε σε μια τελείωτη δίνη λεπτομεριών όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχής και κάθε μέρα δουλεύουμε με κράτη-μέλη και περιφέρειες ε, επί των προγραμμάτων. Όταν κάτι δεν καλύπτεται ρητός ε, στους κανονισμούς, φταίει η Κομισιόν που δεν το συμπεριέλαβε. Όταν κάτι υπάρχει στον κανονισμό και δεν είναι αρκετά σαφές, ε, πρέπει να υπάρχει κάποια καθοδήγηση. Αλλά αν δώσει η Κομισιόν καθοδήγηση, δεν μας αρέσει αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν, ή είναι πολύ λεπτομερή. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι ό,τι και αν υπάρχει με στον κανονισμό, όσο και αν νομίζουμε ότι είναι σαφές, πάντα επιδέχεται ερμηνείας. Να σας δώσω δύο παραδείγματα έτσι τα γρήγορα. Υπάρχει ένα παράρτημα στον κανονισμό κοινών διατάξεων για τα μέτρα δημοσιότητας. Και αυτό αφορά τους δικαιούχους. Είναι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για τη δημοσιότητα. Μπορούμε να συζητήσουμε αν χρειάζονται τέτοιοι κανόνες δημοσιότητας, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οπότε το παράρτημα μιλάει για τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν οι δικαιούχοι. Λάβαμε λοιπόν ερώτημα από ένα κράτος μέλος που λέει αυτά ισχύουν ε, για κάποιους ε, οι οποίοι ε, δεν έχουν ακόμα επιλεγεί ως δικαιούχοι. Αυτό πέρασε μέσα από ένα ολόκληρο κράτος μέλος και κανείς δεν είπε ότι «Ο βεβαίως όχι γιατί δεν είναι δικαιούχοι». Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα, δεύτερο, υπήρχε μια διάταξη στον κανονισμό για τις επιτροπές παρακολούθησης ε, για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που λέει πως ε, θα δημοσιεύει το κατάλογο ε, των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και ένα πρόγραμμα μας ρώτησε αυτό σημαίνει πως δημοσιεύουμε τα ονόματα των μελών ή μόνο τον οργανισμό που εκπροσωπούν. Και πάλι δηλαδή αυτό πέρασε μια ολόκληρη διοίκηση ενός κράτους μέλους κάποιο Υπουργείο και κανείς δεν είπε «Ε, «Μα δημοσιεύστε τα ονόματα, αυτά είναι τα μέλη». Όλα αυτά έρχονται στην Κομισιόν και σας δίνω δύο απλά παραδείγματα. Οπότε τα στρώματα, το επίπεδο ερμηνείας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ περιπλοκό. Πριν φτάσουμε στις δύσκολες ερωτήσεις, στις οποίες ούτε εμείς ξέρουμε την απάντηση. Νομίζω λοιπόν πως ε, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά για το πώς αντιμετωπίζουμε την απλοποίηση. Γι' αυτό ακριβώς η κυρία Κρέτσου συνέστησε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση ε, των δικαιούχων και θέλαμε βεβαίως ε, Καλός ανθρώπου εκεί πέρα, γι' αυτό ακριβώς είναι και ο κύριος που κάθε δίπλα μου μέλος αυτής τη ομάδας. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα αυτή δημοσίευσε τα πρώτα τη ε, συμπεράσματα, τα οποία ελπίζω να έχετε ήδη λάβει από την Κομισιόν και αυτά είναι επίσης διαθέσιμα στο site της ομάδας υψηλού επίπεδου και τα συμπεράσματα αυτά νομίζω ταιριάζουν πολύ με τις συζητήσεις που κάνουμε σήμερα γιατί αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική συνοχή και το απλοποιημένο κόστος. Και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει η ομάδα είναι να δει δύο τομείς πιθανότητων ταυτόχρονα. Εξετάζουν τις ευρύτερες ε, μέσω μακροπρόθεσμες πολιτικές για το πώς θα αναπτύξουμε νέες ιδέες και για το απλοποιημένο κόστος και για την πολιτική συνοχή και ειδικά όσον αφορά την απλοποίηση του κόστους υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συστάσεις προς την Κομισιόν για το τι πρέπει να αλλάξει και ακούσατε κάποια από αυτά τα στοιχεία ήδη σήμερα που μιλάει για περισσότερα ποσά καταποκοπήν, για απλοποίηση της χρήσης για την ε, σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν είναι το πώς θα αντιδράσουμε ειδικά σε σχέση με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και την ε, επανεξέτασή του. Και θα πρέπει ήδη από αυτή την περίοδο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για να ε, έχουμε κάνει τη διαφορά το 2014. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο σε εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, ξέρουμε πως οργανώσατε μία σειρά σεμιναρίων. Να μας ενημερώσετε λίγο για τις δραστηριότητές σας. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή ε, των Περιφερειών θα έπρεπε να εκπροσωπείτε από έναν ε, συνάδελφο, ο Πέτερ Όσφαλτ, ε, θα... που είναι και αρμόδιος για την απλούστευση, θα έρθει αργότερα, αλλά θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία τα δύο εργαστήρια ε, με την ομάδα εργασία του Συμβουλίου Ολλανδικής Προεδρίας και σε συνεργασία με την Ολλανδική Προεδρία βέβαια και το, την Επιτροπή των Περιφερειών. Δύο ήταν τα θέματα. Τι μπορούμε να κάνουμε βράχη πρόθεσμα και τι μπορούμε να κάνουμε μάκρο πρόθεσμα. Αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε να απαντήσουμε. Το ecohesion ήταν ένα ζήτημα. Είχαμε 100 συμμετέχοντες σε αυτά τα δύο εργαστήρια, στο καθένα δηλαδή. 45 feedback, γραπτές συνεισφορές και θα σας πω για το βραχυπρόσωπο και για το μακροπρόθεσμο κάποια από αυτά ε, τα σχόλια που πήραμε, όχι σε επίσημη θέση, απλά ως feedback. Καλό θα ήταν πιστεύουμε να σας ενημερώσουμε για το τι λέτε. Σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταχείριση υπήρχε ένα πρόβλημα είπαν κάποιοι. Σε ό,τι αφορά και το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής συνοχής και άλλα. Δηλαδή, αν έχει πάρει από το πρόγραμμα Horizon ε, μια επιδότηση, ε, μια ΜΜΕ, δεν εντάσσεται στις κρατικές ενισχύσεις. Αν όμως ακριβώς η ίδια επιδότηση δοθεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, εκεί υπόκειται στις κρατικές ενισχύσεις, άρα υπάρχουν ασυνέπειες εδώ. Σαν από τα εργαστήρια ακούστηκε η πρόταση να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κάποιου είδους ε, γενικής εξαίρεσης και για την πολιτική συνοχή ό,τι αφορά τι κρατικέ ενισχύσει και ιδίω για του τομεί όπου υπάρχει διασύνδεση μεταξύ στόχου ε, τη ευρωπαϊκή πολιτική και συγκεκριμένου ε, προγράμματο. Ο έλεγχο επίση, ο λογιστικό είναι ένα θέμα. Εάν θέλουμε να βασιστούμε σε επιδόσει, δεν έχουμε μεγάλη χρήση ε, ε, και απορροφησιμότητα των προγραμμάτων. Πώς θα το εκτιμήσουν αυτό οι ελεκτέ εκ των υστέρων. Είναι πολύ σημαντικό και είναι μια σύσταση που ακούστηκε να δοθούμε εξωτερές διευκρινήσει στην αρχή. Να είναι πιο ξεκάθαρο για όλου του ελεκτές και σε όλα τα επίπεδα ελέγχου ε, να του εξηγήσουν πώ θα το βλέπουν αυτό όταν κάνουν του ελέγχου. Γιατί τελικά βλέπουμε ότι γίνεται κατανοητό διαφορετικά και υπάρχει θέμα για το δικαιούχο αυτομάτως. Έπειτα ένα άλλο θέμα ήταν η μείωση των απαιτήσεων για τις απαιτήσει αναφοράς για, για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και υπάρχουν και προτάσεις κομισιών για καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα για το μακροπρόθεσμο επίπεδο. Φυσικά και πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα σε βάθος από τη Δημοσιονομική Αρχή, από το ελεκτικό για το πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε με βάση περισσότερο την παραγωγή, το output και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις υποχρεώσεις. Και υπάρχει και το ζήτημα βέβαια του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. Απλούστευση μπορούμε να έχουμε μόνο με απλούστερους κανόνες. Και βέβαια και περισσότερη αναλογικότητα. Αυτά προέκυψαν από αυτή τη συζήτηση. Για την ηλεκτρονική συνοχή, το EcoHusion σχετίζεται με τη διοικητική πολυπλοκότητα. Αν δεν μειωθεί αυτή, δεν μπορεί να βοηθήσει και το οικοχίζου. Επανεπιβεβαιώνω δηλαδή αυτά που είπατε κι εσείς νωρίτερα. Θα συντάξω μαζί με την Προεδρία μια έκθεση και θα την ε, υποβάλουμε στην Κομισιόν στα τέλη του μήνα θα ενταχθεί και στη γνωμοδότησή μας για την ε, απλούστευση. απλούστευση. Είναι μια γνωμοδότηση του Πέτερ Όσβαλ, την οποία θα έχει έτοιμη αργότερα φέτος και βέβαια να επανέλθουμε ευχαρίστως εδώ για να σας αναφέρουμε σε πολιτικό επίπεδο τα πορίσματά μας. Θα συνεχίσουμε και επί Σλοβακικής Προεδρίας και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, ιδίω διότι Υπάρχει μεγάλη ανάγκη απλούστευση και στην εδαφική συνεργασία, ιδίω ε, με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στι διασυνοριακέ συνεργασίε. Θα εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, αργότερα θα έχουμε σχετική δράση και θα λάβουμε υπόψη μα ε, ε, το feedback το οποίο σας το μεταφέρουμε σε εσά η Επιτροπή σας εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε όλες τις απόψεις από τις εμπειρογνώμονες Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειών, σχόλια από τους συναδέλφους. Κύριε Μπρέσο. Ευχαριστώ καταρχάς για την προσπάθεια που κάνατε όλοι εκεί. Λυπούμε που είστε πίσω μου και δεν μπορώ να γυρίσω να σας μιλώ. Ευχαριστώ πάντως όλους σας για τις προσπάθειες που κάνατε για να μας παρουσιάσετε την άποψή σας για αυτό το σύνθετο ζήτημα. Προς την Κομισιόν έχω μία ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τι σκέφτονται οι άλλοι. Όπως έγινε και με τους κανόνες ε, για τον ανταγωνισμό, θα το θυμάστε κάποιοι, στο παρελθόν πολλά προϊόντα που πολλούνταν από τη μία χώρα στην άλλη δεσμεύονταν από τη χώρα στην οποία ήθελαν να απολυθούν γιατί εφαρμοζόντουσαν διαφορετικοί κανόνες. Κάθε χώρα εφάρμοζε διαφορετικούς κανόνες υγειονομικού, ασφάλειας ε, κτλ. Εν τέλει, μια ιστορική απόφαση του δικαστηρίου έφερε, αποφάσισε ότι ένα Ολλανδικό προϊόν ε, που, πολλού, που επολύτω ελεύθερα στην Ολλανδία θα μπορούσε να ε, πολιθεί και στη Βουλγαρία διότι υπήρξε ε, ομοιογενής αντιμετώπιση των κανόνων και εφαρμογή των κανόνων στην Ευρώπη. Δεν μπορούσε μια χώρα δηλαδή της Ευρώπης να εφαρμόζει, να μην επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων που γινόντουσαν σε άλλη. Το ίδιο γίνεται και με την λογιστική των χωρών. Ζητήθηκε από τα κράτη να έχουν κοινού κανόνες λογιστικής απεικόνησης. Όλες οι διοικήσεις, οι εθνικές διοικήσεις εφαρμόζουν κανόνες λογιστικής απεικόνησης που συμμορφώνται όλο και περισσότερο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όσο συμβαίνει αυτό, γιατί τέλος πάντων πρέπει να ζητάμε περαιτέρω απολογισμούς με διαφορετικούς κανόνες. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να σέβεται τους δικούς του εθνικούς κανόνες ε, λογιστικής απεικόνησης που έγιναν ομοιογενείς και ακολουθούν τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι από την όλα τις εθνικές αρχές αν το θέλει, γίνονται εκ των υστέρων έλεγχοι. Θα έπρεπε λοιπόν να ξεπεράσουμε την λογιστική απόδοση που εξασφαλίζεται με βάση τους κανόνες κάθε χώρας και άρα απλοποιώντας τεράστια διότι δεν πρέπει να κάνουμε χωριστή διαφοροποιημένη λογιστική επικόνηση μετά το οποίο αυτό που θα έπρεπε να εξεταστεί υλοποιείται. Δηλαδή διαπιστώνεται αν αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Είναι εκεί αυτό το έργο. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε προς την κατεύθυνση εκείνη, γιατί κάθε φορά για να προποιήσουμε υιοθετούμε νέους κανόνες. Όπως κάναμε για τον ανταγωνισμό, λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να πωλήσουμε εκτός χωρών τα προϊόντα μιας χώρας είναι να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βάσει των κανόνων που ισχύουν εξάντε. Αυτό ισχύει και για τα, για τα λογιστικά. Να πάμε προς την κατεύθυνση εκεί κάνοντας μια ριζοσπαστική, δραστική μείωση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι έχω έξι βουλευτές που θα λάβουν το λόγο. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι λοιπόν. Ένα με δύο λεπτά. Κύριε λέω, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Και το 7 είναι, ξέρετε, ιερός αριθμός. Χαίρομαι που έχουμε τόσους ομιλητές. Λοιπόν, Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η πρόοδος για την ε, επιλογή απλοποιημένου κόστους, οπότε σημειώνεται πρόοδος, δεν υπάρχει μόνο κριτική. Ένα άλλο θέμα είναι ότι σκοπεύαμε να πούμε ότι εντάξει, ε, θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά μια θεματική εστίαση, μια αιρεσιμότητα εξάντε για να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα. Έχουμε το πρώτο έτος ε, που βεβαίως ε, τα πράγματα ξεκινάνε πάρα πολύ δύσκολα και θα έλεγα ότι είμαστε στο πρώτο 15 λεπτό ενός ποδοσφαιρικού αγώνα οπότε θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο έχουμε βάλει κατά μέρος 20 δισεκατομμύρια για αυτούς οι οποίοι όντως θα αποδώσουν οπότε κανείς δεν μίλησε ακριβώ για αυτή την φάση που είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν αυτές τις συμφωνίες εταιρικής ε, σχέσης για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα και κανείς δεν το σχολίασε. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά ακριβώς την εμπιστοσύνη και τον ε, έλεγχο και δεν ξέρω. Ακούγοντας την Κομισιόν απελπίστηκα. Γιατί τώρα αυτή η πολιτική ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια. Και οι εισηγητέ λένε ότι έχουμε τον κανονισμό και κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει, λέτε ότι σας ρωτάνε διάφορα εξωτερικά πράγματα. Μα πού είναι το λάθος. Κάναμε τα σωστά πράγματα στον κανονισμό. Και τι μπορεί να αλλάξει εύκολα, γιατί η Κομισιόν λέει πως θα έπρεπε να υπάρχει ήδη μια απλοποίηση. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Μιλάμε για το Εράσμους και τα άλλα προγράμματα για τον ορίζοντα 2020 κτλ. Εγώ θεωρώ ότι η απλοποίηση εκεί, π.χ. στον ορίζοντα 2020, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε γιατί ε, εκεί πέρα ακούμε πάρα πολύ θετικά πράγματα για το πώς το βλέπουν ε, οι δικαιούχοι. Οπότε, το να μαθαίνουμε δεν σημαίνει απλά να κινούμαστε όλοι στον ίδιο χώρο, αλλά να κοιτάμε και παρά έξω. Κοιτάξατε άλλες ε, πολιτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Ρόπε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Το θέμα μας είναι πολύ σύνθετο και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα. Αυτοί που πρέπει να εφαρμόζουν τις διαδικασίες έχουν, αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα. Εγώ όταν ήμουν στο Δήμο είχα ασχοληθεί με αιτήσει και έχω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, τα διαφορετικά, τα, το, τα ταμεία ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Αυτό δυσχεραίνει πολύ τη ζωή των ετούντων αλλά και των επιτροπών ε, και οργάνων παρακολούθησης. Ίσως θα έπρεπε να μιλάμε όχι για απλοποίηση αλλά για βελτίωση των κανόνων. Δεν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να έρθει η ο σωστός χρόνος, αλλά να βελτιώσουμε αμέσως το σύστημα, κάνοντάς το καλύτερο. Όταν δημιουργείται νέο ταμείο, δημιουργούνται νέοι κανόνες. Και ο καθένας χάνει χρόνο προσπαθώντας να καταλάβει τι λένε. Αυτό είναι απώλεια και χρόνου και χρήματος. Η διαδικασία θα έπρεπε λοιπόν να είναι σαφής όσο καλύτερη γίνεται. Θα έπρεπε να αποφύγουμε ελέγχους επιπρόσθετους. Γιατί όσο πιο ορθολογική είναι η διοίκηση, τόσο περισσότεροι πόροι υπάρχουν για να κάνουμε πράγματα. Η απλοποίηση θα μειώσει και το διοικητικό βάρος και θα μας επιτρέψει να έχουμε υψηλότερη ποιότητα με μικρότερο κόστος. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσον θα μπορούμε να πετύχουμε την προσθέμενη αξία που θέλουμε. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάποια κράτη-μέλη κάποιες φορές για να αποφύγουν προβλήματα αρχίζουν να ασχολούνται με την αύξηση του νομοθετικού ε, της νομοθετικής και κανονιστικής επιβάρυνσης χωρίς δικαιολογία. Κάτι άλλο σημαντικό στον τομέα της απλοποίησης είναι η ανάγκη να απλοποιηθούν οι οδηγοί. Δεν είναι σημαντικό να απλοποιούμε μόνο ε, τα νομοθετικά κείμενα, αλλά και την εφαρμογή τους. Η Επιτροπή αυτή αυτή έχει δώσει, έχει θέσει τον στόχο της απλοποίησης. Με εκπλήσει λοιπόν όταν έχει η Κομισιόν και λέει μην περιμένετε πολλά πράγματα από όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι η καθήκον της Επιτροπής να βελτιώσει τα νομικά κείμενα για να πετύχει αποτελέσματα και να βελτιώσει την κατάσταση συνολικά. Ευχαριστώ. κύριος Ρούλαντ, έχει το λόγο. Ναι, δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διάφορους ε, ομιλητές Συμφωνώ με την κυρία Μοχό που μίλησε πριν από λίγο ε, και να σας μεταφέρω μια μαρτυρία και μετά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ως δήμαρχος καταρχάς μιας μικρής, ε, ενός μικρού γαλλικού δήμου από το Λίγυρα να σας πω ότι ε, ακούμε και το ξέρουμε βέβαια, αλλά ακούμε ότι τους αποθαρρύνει το υπερβολικό κόστος, τα, τα δικαιολογητικά, προθεσμίες για τις κτλ. Επί τόπου δίνεται κακή εικόνα τελικά, ε, λόγω ακριβώς αυτής της πολυπλοκότητας. Σε ό,τι αφορά την ουσία τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε μόνο μία ιδέα, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά την απλούστευση Ρεαλιστέ Αυτό θα πει καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστούν από κοινού και να μην πέσουν στον πειρασμό ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ασφάλματα γιατί αυτό δεν λύνει το πρόβλημα οι δικαιούχοι ε, αυτό που θέλουν είναι πρόοδος επιτόπου και τα κράτη, η ε, Κομισιόν από κοινού πρέπει να προχωρήσουν να προοδεύσουν. Μια άλλη παρατήρηση, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές πάντα, θα πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, ιδίω ε, και ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχει και αυτό μερίδιο ευθυνών για την πολυπλοκότητα που σήμερα καταγγέλουμε. Τρίτο σημείο. Για να είμαστε πάντα ρεαλιστές πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι είναι επίγον ε, επειδή πολλοί δικαιούχοι λένε ε, ε, δεν στρέφονται πλέον στην πολιτική συνοχή. Έχουμε την απόφαση των Βρετανών σύντομα. Έχουμε τα πολύ ψηλά ποσοστά των ευρωσκεπτικιστών σε διάφορες χώρες. Και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, όπως και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα διοικητικά προβλήματα και η υποεκμετάλλευση των κονδυλίων ε, συνεπάγεται και ε, πρόβλημα με την αξιοπιστία μας. Άρα πρέπει ε, να είμαστε ρεαλιστές. Και τελειώνω, να είμαστε ρεαλιστές και σε ό,τι αφορά τη μέθοδο. Δηλαδή η Κομισιό, το Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε ποια είναι τα αποτελεσματικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν τάχιστα, χωρίς να χρειαστεί να νομοθετήσουμε εκ νέου και να γίνει διάκριση μεταξύ του τι μπορεί να περιμένει μέχρι το 2020 και το τι είναι άμεσο να γίνει. Γιατί θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό το να αλλάξουμε άρνητα πράγματα σε διαφορά το κόστος. Αλλά σίγουρα κάποιες τροποποίησεις πρέπει να γίνουν μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. κυρία Λέτιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας για την πολύ καλή, τις πολύ καλές παρουσιάσεις και για το ότι βεβαίως μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας μαζί μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι άλλαξε η πολιτική συνοχής από τη μία περίοδο χρηματοδότηση στην επόμενη και τώρα καταλήξαμε βεβαίω με προπολογισμό ο οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα αλλά κοιτάζοντα τα συστήματα ελέγχου και δημοσιονομικού ελέγχου εξακολουθούμε να κοιτάμε το πραγματικό κόστος και επιπλέον και τα αποτελέσματα και την απόδοση. Οπότε κατά βάση δεν παραλείπουμε τίποτα και συνεχώς συσσωρεύουμε στρώματα Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβλήματα με την απλοποίηση γιατί το σύστημα πλέον δεν απλοποιείται αλλά ε, όλο πιο πολύπλοκο γίνεται. Οπότε ελέγχουμε τα πάντα πλέον. Οπότε χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση οπωσδήποτε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά και η Κομισιόν να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να πει στα κράτη-μέλη να μην φοβούνται να χρησιμοποιούν τις, ε, αυτές, τις επιλογές απλοποιημένου κόστους γιατί πρέπει να εστιάζουμε στα αποτελέσματα και όχι μόνο στο πραγματικό κόστος. Γιατί βεβαίως ο τελικός δικαιούχος μπορεί να καθορίσει διαφορετικά το μείγμα κόστους με το οποίο θα επιτύχει το αποτέλεσμα, αλλά εμείς πρέπει να ελέγχουμε τα αποτελέσματα. Και κάτι άλλο το οποίο σχετίζεται και επειδή το αναφέρατε, ε, η διαφορετική αυτή προσέγγιση και το πώς ε, οι διοικήσεις φοβούνται το τι θα πούν οι ελεγκτές. να δοθεί μια συγκεκριμένη οδηγία σε τελικό δικαιούχο. Εμείς είχαμε συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα μας όπου η διοίκηση είπε πράγματα συγκεκριμένα να κάνει στο δικαιούχο. Μετά ήρθαν οι ελεγκτές είπαν ότι ήταν λάθος και τώρα που τα λεφτά έχουν... Τώρα τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν. ποιος ανέλαβε λοιπόν τον κίνδυνο και ποιος φταίει ο τελικός δικαιούχος ο οποίος πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Γιατί δεν μπορεί ε, όλο τον κίνδυνο να τον έχει ο τελικός δικαιούχος. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα ρίσκο στο επίπεδο της διοίκησης. Ακριβώ λόγω της διαφορετικής προσέγγισης μεταξύ των διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τσίλερ, ναι, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα χωρίς κανόνες δεν γίνεται. Έχουμε τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογουμένου ο οποίος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ε, το πώς εξοδεύονται τα λεφτά του και ότι αυτά εξοδεύονται ε, σύμφωνα με τους κανόνες και ότι υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Αυτό δεν γίνεται χωρίς κανόνες. Το θέμα βεβαίως τώρα είναι πόσους κανόνες χρειαζόμαστε και πώς ε, τους εφαρμόζουμε. Στην διαδικασία απαλλαγής ε, διαπιστώσαμε ότι στην εφαρμογή των ε, ταμείων συνοχής έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος 6% το οποίο είναι πολύ πιο πάνω από αυτό το που είχαμε ορίσει ως αποδεκτό όριο το 2% βεβαίως 2 τρίτα των λαθών αυτών είναι λάθη στην προκήρυξη και ως κάποιος ο οποίος ε, είχα σχέση με τις προκηρύξεις μπορώ να πω πως τι έγινε, ήταν κάτι το οποίο έγινε σκεμμένο για να δοθεί σε συγκεκριμένους ε, αναδόχους ή προμηθευτές από την, περιφέρεια, από την ή δεν ήξεραν ε, τους κανόνες. Το πρώτο, η πρώτη περίπτωση είναι σαφώς κατά των κανόνων ανταγωνισμού. Ε, η δεύτερη περίπτωση είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει η διοίκηση να προσέξει να καταρτήσει το προσωπικό της γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις τα κριτήρια αυτά είναι των διαγωνισμών είναι εθνικό δίκτυο ή αν είναι ομοσπονδιακή χώρα όπως η Γερμανία ε, τα κρατήδια έχουν δικό τους δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών. Αν δεν είχαμε λοιπόν αυτά τα δύο τρίτα θα ήμασταν ήδη στο 2%. Ε, βεβαίως μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου σφάλματα. Και βεβαίως πάλι εδώ πέρα οι υπεύθυνοι έγραψαν αυτό το βλιαράκι. Ο Σιμ Κάλλας, ο υπεύθυνος αυτής της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου, μας είπε πως ε, μόνο οι κανονισμοί αυτοί είναι 270 σελίδες. Είναι πάρα πολύ λεπτομερείς. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν άλλες 880 σελίδες της πράξης κατεξιοδότηση μέχρι στιγμή που είναι κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν και την Ομάδα Εργασία του Συμβουλίου. Ε, και αυτό είναι άλλο ένα επιπλέον γραφειοκρατικό στοιχείο. Και μετά λέμε στους ανθρώπους που τα εφαρμόζουν αυτά ότι πρέπει να καταγράφουν τα τηλεφωνήματά τους ε, εάν έγιναν για να γίνει ε, ένα συγκεκριμένο έργο και έχει χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά όχι στην περίπτωση που ήταν ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν αφορούσε αυτή τη δουλειά. Ε, εκεί πέρα πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο τρέλας και πρέπει να παρέμβουμε. Και βεβαίως ε, οι υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται τα κονδύλια είναι οι αρχές του προϋπολογισμού και αν αρχίσουμε να ψαλιδίζουμε τι θα πει ο σκεφτόμενοι το τι θα πει ο ελεγκτής έχουμε ένα αυτόματο φρένο οπότε θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς λειτουργεί και σκέφτεται ο ελεγκτής και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο υπάρχει ήδη η προσέγγιση ότι θέλουμε να κοιτάμε περισσότερο το αποτέλεσμα και όχι τόσο τον τρόπο, ο οποίος πρέπει να είναι σύνομος βεβαίως. Αλλά βεβαίω ε, όταν προσανατολιζόμαστε και στο αποτέλεσμα, όπως σας είπα, εκεί πλέον προσανατολίζεται και το ελεγκτικό συνέδριο και είμαστε όπως είπαμε στην κοινή ε, διαχείριση. Η εποπτεία είναι στις εθνικές αρχές και ελπίζω, όπως είπα, να μην κινούνται οι ελεγκτές με τη σκεπτική ότι εγώ θα ψάχνω μέχρι να βρω ένα σφάλμα. Αλλά έχουμε και τις εφαρμοστικές διατάξεις των διαφόρων ταμείων και θα πρέπει και εκεί πέρα να υπάρχει μία συμβατότητα έτσι ώστε κάποιος ο οποίος ασχολείται με το Περιφερειακό Ταμείο θα μπορεί να διοικεί και κάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Και κάποιος ε, επίσης ο ίδιος να μπορεί να διαχειρίζεται και κάτι το οποίο αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, έχουμε πολλά να κάνουμε. Αυτό είναι αυτό το οποίο ζητάμε μαζί με την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κυρία Νταμάτου. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούμε ότι η απλοποίηση είναι σημαντική. Αυτή, κάνει, αυτή τη δουλειά κάνει η ομάδα μας. Ερωτήσεις για τις υπηρεσίες πληροφορικής. Είναι σωστό πολλά κρατημέλη, περιφέρειες, ιδίω στην Νότια Ευρώπη και στην περιφέρεια γενικότερα, πολλές φορές δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή υποστήριξη για την εφαρμογή μέτρων e-governance όπως ζητούνται. Ρωτώ λοιπόν και από την Επιτροπή και από την ομάδα εργασίας και τους υπαλλήλους που είναι εδώ είναι χρήσιμη να υπάρξει μια μεγαλύτερη βοήθεια προς τις περιοχές αυτές. Άλλη ερώτηση. Μια ειδική μελέτη για τις περιφέρειες εκείνες που ήταν λιγότερο ανεπτυγμένες στην πρώτη περίοδο προγραμματισμού και συνεχίζουν να είναι τώρα. Μετά λένε, γίνεται λόγος για την ανάγκη να μοιραζόμαστε τις βέλτιες πλαστικές τώρα και τις κακές εμπειρίες για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Η ερώτηση που θέτω ωστόσο είναι αυθόρμητη. Καθυστερήσεις. Αναλύουμε λεπτομεριακά κείμενα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε μετά το 2020, αλλά πρέπει να είμαστε έντιμοι μεταξύ μας. Δεν είναι νορμάλ να υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Ιταλία που έχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και όχι μόνο. Τι μέτρα προτείνει η ομάδα για να καλύψει τις, τα εμπόδια της προηγούμενης περίοδου, γιατί αλλιώς ο κίνδυνος είναι να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Απλοποίηση κόστους τώρα. Μιλάμε για αποδεκτές δαπάνες που θα υπολογίζονται με βάση προκαθορισμένη μέθοδο που θα βασίζεται στα αποτελέσματα. Έχετε προτάσεις για να λύσουμε κατάλληλα την αντίφαση μεταξύ μείωσης ε, το, της, γραφει, ε, με ε, ενιαίο συντελεστή πληρωμής ή και τις ε, κρατικές το ίδιο ισχύει και με την έλλειψη διάκρισης μεταξύ σφάλματος και απάτης. Χρειάζονται δηλαδή σαφείς κανόνες για τον έλεγχο ή όχι. Κλείνω ρωτώντας. Προτίθεται να, προτίθεστε να αλλάξετε τους κανονισμούς. Η οχι κλεινω ρωτωντας να υψηλού επίπεδου θα δημιουργήσει και άλλο overlap tipping ή απλώς αλλάζουμε τον κανονισμό ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμασίτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. είναι πολύ λεπτομερείς οι κανόνες και είναι εύκολο να γίνουν σφάλματα, είτε είναι αυτά εσκεμένα είτε όχι. Χρειάζονται απλουστευμένες διαδικασίες ίδιες για όλους, χρειάζεται εναρμόνιση και στην ορολογία, ώστε να μπορούμε να, να μην γίνεται ερμηνεία διαφορετική ή να μην μπορούμε να ερμηνεύουμε όπως μας βολεύει τα πράγματα. Λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών σίγουρα κάποιοι και παρετούνται, εγκαταλείπουν αλλά και κάποιοι κάνουν λάθη. Πρόεδρος να σας υπενθυμίσω ότι τα πρώτα πορίσματα του έργου της ε, ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου σας εστάλησαν από τη γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άρα είστε ενήμεροι πλέον για το έργο της ε, ομάδας ψηλού επίπεδου. Σήμερα Ακούσαμε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμα κατά μισή ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους τους ομιλητές και που συμμετέχονται σε αυτό το εργαστήριο. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Και θα προσπαθήσω τώρα να τηρήσω αυστηρά το χρόνο μέχρι το τέλος της ημέρας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα μέτρα είναι έκθεση της πρωτοβουλίας, η υποφαινόμενη νησυγήτρια και η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η επιτροπή η δική μας. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε συζητήσει τη γενική δομή και την κατεύθυνση της έκθεσής μου πέρυσι το Δεκέμβριο, όμως σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Λίγη ησυχία. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Okay. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Interreg, είναι και ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής. Με πρωταρχικό στόχο να προωθήσει την εναρμόνιση της οικονομικής ε, και εδαφικής ε, ανάπτυξης ένωσης. Το Δεκέμβριο λοιπόν σας υπέβαλα τις βασικές κατευθύνσεις τη γενική δομή του σχεδίου έκθεσής μου. Έλαβα υπόψη τα δικά σας σχόλια και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης ε, πιο λεπτομεριακά, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και παρκή χρόνο στη διάθεσή μας για να το συζητήσουμε. Για την κατάσταση τροπολογιών προτείνω η προθεσμία να είναι Τετάρτη 6 Απριλίου 12 το μεσημέρι για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου. 6 Απριλίου, 24 Μαΐου. 6. 6. Allow me to continue in, in Bulgarian to, to present uh, the, the... Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρά μου να σας ε, παρουσιάζω την έκθεσή μου τους στόχους της ε, πολιτικής ε, συνοχής με κύριο Βάρος την Ευρώπη 2020 και βεβαίως δεύτερο σημείο έμφαση σε την απλοποίηση του Interreg. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, παρά την ε, δική μας την πρόθεση για το να εστιάσουμε στο τωρινό χρονικό πλαίσιο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και υπάρχει τωρινή ε, προγραμματική περίοδος ε, στην οποία θα έπρεπε να δούμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές. Η έκθεσή μας λοιπόν βασίζεται στην έκθεση της ε, Κομισιόν και τις εκθέσεις των κρατών μελών. Και έχουμε και την επέτειο του Ίντερεγκ. Υπάρχει μία δήλωση της ε, Κομισιόν και της Επιτροπής των Περιφερειών υπάρχει επίσης μια ανασκόπηση στην 20 ιστορία του Ίντερεγ και υπάρχουν και συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. και μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις απόψεις των πολιτών που ζουν σε μεθοριακές περιοχές. Υπάρχουν επίσης κάποιες εκθέσεις ε, κλειδί για τις ε, σχετικές ε, περιφέρειες, παραδείγματος χάρη την απλοποίηση της πολιτικής, ε, την συνεργασία μεταξύ περιφερειών κτλ. Παραδείγματος χάρη, για την διασυνοριακή συνεργασία. Τώρα πλέον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ε, και υπάρχει και η μετάβαση προς την καινοτομία και μια μεγαλύτερη εστίαση στις οικολογικές πτυχές και οι διασυνοριακές συνεργασίες. Οι διασυνοριακές συνεργασίες στηρίζουν την ε, οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας και έτσι βελτιώνεται και η διοικητική ικανότητα. Οι περιφέρειες ε, και οι πόλεις ε, ανταλλάσσουν βέλτιστες ε, πρακτικές και έτσι βελτιώνουν τις πρακτικές που ακολουθούν. Έχω αναφέρει συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα στην έκθεσή μου. Επίση, ανεξαρτήτως από το γεγονός ότι το Ίντερεγκ είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής ε, σύνοχης, αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν οι περιορισμοί του προϋπολογισμού, και δεν μπορούμε να πτύχουμε όλους τους στόχους. Κάποια πράγματα εγκρίθηκαν αργά και απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη να αναλάβουν κάποια βήματα για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Η ανταλλαγή δεδομένων για την διασυνοριακή εφαρμογή είναι αναγκαία όλα τα σχετικά όργανα θα πρέπει να χρησιμοποιούν μία ενιαία μέθοδο. Ή δε φορείς ε, θα πρέπει να έχουν μία ενιαία πολιτική όσον αφορά τις εκθέσεις, ε, τις αναφορές, ε, το ίντερνετ εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ε, τυποποίηση. Υπάρχει μια μελέτη του ΕΣΠΟΝ για τα διάφορα σενάρια κατά το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να προγραμματίσουμε την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Υπάρχουν δύο μέσα οι ολοκληρωμένες περιφερειακές επενδύσεις και μια ανάπτυξη, μια εξέλιξη και ανάπτυξη υπό την ηγεσία των Δήμων λειτουργεί νομίζω καλά η συνεργασία και υπάρχουν βεβαίως και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι από μακρισμένες περιφέρειες ε, πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την εδαφική ολοκλήρωση. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μακροπεριφερειών. Επίσης η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί. Όλες οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, ε, υπάρχει μεγάλη μεταναστευτική πίεση και εδώ πέρα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν μιλάμε για κοινοτομία, για κοινοτομία και την διάδοση των βέλτιστων πρακτικών πρέπει να δούμε τις στρατηγικές εξειδίκευσης όπως επίσης και τα δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχουν κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης συνεργασιών και δίκτυα συνεργασιών. Επίσης ζητάμε στην έκθεση την έγκριση διασυνοριακών πρακτικών για την εξειδίκευση. Επίσης σημαντικέ είναι οι ευρωπαϊκές ενώσεις για την διασυνοριακή συνεργασία, η ευελιξία σε σχέση με την πλατφόρμα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και βεβαίως ε, ζητάμε να υπάρξουν τέτοιες ομάδες σε όλες τις χώρες π.χ. μπορούν οι χώρες να παραδειγματιστούν από το Λουξεμβούργο για την ε, σύσταση ευρωπαϊκών συνδέσμων και με τον τρόπο αυτόν ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν επίσης και τις ε, προκλήσεις που σχετίζονται με τα μεταναστευτικά φαινόμενα. Βεβαίω θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και περαιτέρω ευέλικτοι μηχανισμοί σε συνδυασμό με την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει για την περίοδο την προγραμματική 2007-2013 δεν υπήρχαν αρκετές ε, παρατηρήσεις ε, για τα προγράμματα εδαφικής ε, συνεργασίας. Υπάρχουν διάφορα τέτοια μέσα. Υπάρχουν, όπως είπα, και οι δυνατότητες ε, του ΕΦΣΙ, του προγράμματος Juncker και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων. Ανεξαρτήτως λοιπόν από την ύπαρξη του κανονισμού του Interreg ε, εξακολουθεί η χρήση του να είναι πάρα πολύ δύσκολη πρέπει και εδώ πέρα να υπάρξει κάποια απλοποίηση. και των ε, κανόνων. Ποιες συστάσεις έχουμε τώρα για το μέλλον. Περιφερειακή και τοπική συνεργασία έχει αποδείξει την σημασία της το Interreg πρέπει να διατηρηθεί ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και πρέπει να, λάβει μεγαλύτερο, να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο για τον σχεδιασμό της πολιτικής μετά το 2020. Συνολικά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην διασυνοριακή συνεργασία. Τα προγράμματα δεν ναι, θα πρέπει να μοιράζονται μόνο με βάση τον πληθυσμό αλλά να ισχύσουν και κάποια άλλα κριτήρια. Χρειάζονται ειδικές στρατηγικές για τις μεθοριακές περιοχές για να υπάρχει μια διαρκής και σταθερή ανάπτυξη. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και η παραπέρα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίση, η πρόταση της Προεδρίας του Λουξεμβούργου πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη και με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών να προγραμματιστούν νέα βήματα το 2016 θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μέλλον του Interreg μετά το 2020 πάντα σε σχέση με την ε, προετοιμασία της πολιτικής ε, περιφερειακής ε, ανάπτυξης. Εδώ πέρα λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε τα αποτελέσματα των ε, ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εδώ πρέπει όλα όλοι οι σχετικοί φορείς να έχουν κάποιες ολοκληρωμένες πλατφόρμες για να ενημερώνονται οι χρήστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην έκθεσή μου και αναμένω την αντίδραση των συναδέλφων και των ειδικών και από κοινού μπορούμε νομίζω να γράψουμε μια έκθεση η οποία θα ενσωματώνει τα σημαντικότερα στοιχεία. yes. Αυτή ήταν η παρουσίαση της έκθεσης και τώρα δίνω το λόγο στους και ηγητές. Η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η εδαφική συνοχή είναι κλειδί της, του στόχου ανάπτυξης της Ένωσης στο εδαφικό τομέα, γιατί μέσω αυτού επιτρέπεται η συνεργασία για τον εντοπισμό κοινών λύσεων σε, περιοχή, σε θέματα όπως ε, την ανάπτυξη υπέρθου, τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, τη δημιουργία μικρομεσαίων, δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η, τα δίκτυα μεταφορών, η περιβαλλοντική ε, πολιτική, η ανάπτυξη, η έρευνα είναι παραδείγματα άλλων τομέων που αναδεικνύουν την προτεραιότητα αυτή. Ταυτόχρονα οι διάφορες περιοχές της Ένωσης μπορεί να συνεργαστούν με άλλες περιφέρειες σε κοινά έργα για την μείωση του, των διασυνοριακών επιπτώσεων. Ο εντοπισμός των περιοχών με τις μεγαλύτερες και πιεστικότερες ανάγκες είναι πολύ σημαντικό, όπως και να εμπλέκουμε τις τοπικές αρχές και την δομή, τα στάνταρ αξιολόγησης και διαβούλευσης που οδήγησαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και τη δημιουργία ενός ενιαίου πολυεπιπέδου συστήματος διακυβέρνησης. Μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία αυτή δίνει την ευκαιρία σε όλους οπουδήποτε στην Ευρώπη να μετάσχουν στην κοινή αγορά και να κερδίσουν από τα πλονεκτήματα αυτά. Η πολιτική συνοχή, η εδαφική συνεργασία δηλαδή, αντιπροσωπεύει την ορατή πλευρά της ενιαίας αγοράς που έχουν στόχο να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, οικονομική άνοδο της Ένωσης βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονομιών. Αυτό βοηθά να παράσχουμε ευρωπαϊκά προϊόντα που η αγορά δεν μπορεί να προμηθεύσει. Κάθε ευρωπαϊκό έδαφος έχει το δικό του ρόλο και πρέπει να γίνει πηγή ανάπτυξης αυτή καθεαυτή μέσω δίκαιης κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η πρόσφατη οικονομική ανάλυση επιβεβαίωσε την προσέγγιση αυτή μέσω πολλών ερευνών που αποδεικνύουν ότι η γεωγραφία μετράει. Η περιφερειακή πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η εδαφική συνεργασία αποτελεί επίσης το απαραίτητο πλαίσιο για την εμπλοκή εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών στις θεμελιώδεις στρατηγικές και στην δημιουργία δικτύων που ξεπερνούν τα φυσικά και πολιτικά όρια των χωρών. παρότι δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για το πώς αναπτύσσονται αυτές οι συνεργασίες, κάποιες αρχές όπως η διαφάνεια, η επικουρικότητα, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η λογοδοσία ε, συνυπάρχουν. Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού ε, τομέα θα διευκολύνει την αποκέντρωση και την εμπλοκή συμμετοχή όλης της κοινωνίας. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να προσαρμοστούν στις πιέσεις της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η αλλαγή του κλίματος συνιστά απειλή για πολλούς κλάδους, ενώ είναι ευκαιρία για άλλους. Οι δημοκρατικέ αλλαγέ και η γύρανση του πληθυσμού απαιτούν νέε πολιτικές στην αγορά εργασία. Και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις οικονομικές αλλαγές απαιτήσουν νέες προσεγγίσεις. Ενώ όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδοκίες, πρέπει να έχει και μια σωστή πολιτική συνοχής για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ε, ένα από τα θέματα που όλοι επιδιώκουμε είναι η κοινή πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε η Ένωση να έχει τα αναγκαία μέσα για ανάπτυξη και βιώσιμη οικονομική ε, μεγέθυνση. Άλλωστε οι πόλεις και οι περιφέρειες εφαρμόζουν μέτρα και ε, κοινοτικά που υλοποιούν και την κοινοτική νομοθεσία. Δεν πρέπει λοιπόν να παρακολουθούν απαθώς, αλλά να εμπλέκονται ως πραγματικοί ε, εταίροι στις διαδικασίες αυτές. Ευχαριστώ. Άλλη σκιώδης τώρα. Ρόπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήμουν δήμαρχος σε μια πόλη στη Λεθανική Μεθόριο. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Μιχαηλόβα για την έκθεση που συνέταξε. Η συνεργασία και η διασυνορική συνεργασία είναι θετικός παράγοντας, είναι σχετικός παράγοντας. Βέβαια πρέπει να εκφράσω την ανησυχία μου σε ό,τι αφορά τον πάρα πολύ ε, λίγο προϋπολογισμό. Περιμένουμε η Κομισιό να προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα, διότι θέλουμε έγκαιρα να εφαρμοστούν τα μέτρα όπως και η απλούστευση των κανόνων για τα διάφορα έργα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης τώρα, έχω κάποιες ε, ανησυχίες, παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά τον ειδικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Σίγουρα η χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ είναι θετική, είναι ευεργετική, αλλά χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς δηλαδή βλέπετε το ρόλο της τράπεζας στο πλαίσιο της ενταφικής συνεργασίας. Νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να δίνει έμφαση στις αποκεντρωτικές τάσεις ε, της ενταφικής συνεργασίας. Πολλές δράσεις αποσκοπούν ε, στο να βοηθήσουν μεθορικές περιοχές, αλλά Πολλές φορές η διαχείριση γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, από το κέντρο δηλαδή και όχι στην περιφέρεια. Οι περιφέρειες δεν έχουν τους ειδικού που έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες. Δεν έχουμε ταμείο που να χρηματοδοτεί επίσης μικρής κλίμακας έργα. Αλλά αυτό θα ήταν ένα καλό μέτρο για την ε, βελτίωση των διοικητικών μας δυνατοτήτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε μήπως ε, οι δαφικές επενδύσεις θα μπορούσαν ε, να προωθηθούν. Και σε ό,τι αφορά τα σύνορα, πρέπει να γίνουν πιο κοντά, πιο πολλά κοντά στα σύνορα, σε μεθορικές περιοχές. Υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούν καταστάσεις επίγοντος σε μεθορικές περιοχές όπως είναι σήμερα η προσφυγική κρίση. Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με τις απαιτούμενες επενδύσεις. Έχουμε αυτές τις 11 προτεραιότητες, αλλά σωστά επιβάλλει αυτές τις απαιτήσεις η Κομισιόν. Θα έπρεπε ίσως η Κομισιόν να δει κατά πόσο η θεματική συγκέντρωση ήταν ή όχι ευεργετική τελικά. Ο κύριος Φανίστελ Ρόιλ, η πρόεδρος, εκ μέρου ε, του Σκιώδου, αν πάρετε το λόγο. Ναι, ο κύριος ε, Χέκμαρκ δεν μπορεί να είναι εδώ. Αλλά είναι απλό το μήνυμα που θέλουμε να σας ε, παρουσιάσουμε. Θεωρούμε ότι η έκθεση είναι πολύ καλή, πολύ πλήρης. Είναι πολύ καλή η έκθεσή σας. τέσσερις ε, τομείς, ε, τα είπαμε και πιο πριν, απλούστευση. Ίσως ε, οι εξωτερικές, τα εξωτερικά σύνορα, αυτές οι σκέψεις που ακούσαμε και από τον προλαλήσαντα. Γιατί έχει να κάνει και με τον κανονισμό, με την αξιολόγηση επιδόσεων κτλ. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα δαυκής συνεργασίας. Ε, μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες την προστέμενη ευρωπαϊκή αξία. Στην έκθεσή σας υπάρχει και ένα κεφάλαιο για το μέλλον. Θα μπορούσαμε ίσως εδώ να προσθέσουμε κάτι, τονίζοντας τη σχέση μεταξύ εδαφικής σύνοχης, φυσικά σε αυτήν, και εδαφικής συνεργασίας, που είναι το κείμενο αυτής της έκθεσης. Και ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για τη συνθήκη και να συνδέσουμε γιατί έχουμε την κοινωνική, οικονομική και την εδαφική συνοχή. Και αυτό το τρίτο σκέλος είναι, είναι και αυτό σημαντικό. Όταν έχουμε λοιπόν νέε συζητήσεις για τα ταμεία και για τη χρηματοδότηση και για τις αποζημιώσεις, θα πρέπει να δούμε αν η πολιτική στόχο έχει την τόνωση της καινοτομίας. Βιωσιμότητα, ΜΜΕ, κοινωνικές πτυχές επίσης είναι σημαντικές. Να πω και κάτι ακόμη. Τι έκανε η Κομισιόν. Τίποτα δεν έκανε επί της ουσίας. Εμείς το κάνουμε στο Κοινοβούλιο και είπαμε ότι θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εδαφική διάσταση. Άρα θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε στην έκθεση αυτό. Και τώρα αν σκεφτείτε πιο πέρα και πιο μακριά και δείτε τι συνιστά προσθέμενη αξία. Τα διασυνορικά, μακροπεριφέρειες, συνεργασία σε αυτό το επίπεδο στις μεθορικές περιοχές είναι που η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει περισσότερο παρά στο 2,8% του προϋπολογισμού συνοχής. Αν δαπανίσουμε το 50% των κοντιλίων συνοχής στην εδαφική συνεργασία και στα σχετικά εργαλεία, μπορεί και να έχουμε μια απόλυτη προσταμένη αξία. Κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερη σε σχέση με τα εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Επίσης, αν ε, μιλήσετε με τους συναδέλφους σας, στις ομάδες σας ε, και ε, στα Εθνικά Κοινοβουλία θα σας πούνε δευκή συνεργασία είναι σημαντική, κάτι που θα σας πούνε η περιφερειακή πολιτική είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε επίπεδο κρατών μελών. Η διασυνοριακή πολιτική είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Και ισχύει αυτό βέβαια και για τα νησιά. Θα πρέπει να προωθήσουμε ειδικέ εδαφικές θέσεις. Να δούμε τώρα τι τροπολίες μπορούμε να καταθέσουμε. Εγώ τι προσδοκώ και για τους πολίτες μας και για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τους άλλους στο Κοινοβούλιο, να εξηγήσουμε ότι η ενταφική συνεργασία πρέπει να έχει ένα πιο προβεβλημένο ρόλο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Άρα στο τελευταίο τμήμα που μιλάτε για το μέλλον σκεφτείτε το. Μήπως μπορείτε να το συμπεριλάβετε. Μπορούσα να το λάβω και εγώ υπόψη στη δική μου την έκθεση, εάν περάσει εδώ. Ευχαριστώ. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ. Τόμασιτς. Για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ. Ε, λείπει ο συνάδελφος ε, γιατί θέλει να πάει την πήγε στην εκλογική του περιφέρεια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και πρόεδρο για μια εξαιρετική έκθεση και πολύ καλές προτάσεις που κάνει. Οι περιφερειακές, οι ακραίες ε, συνοριακές περιοχές της Ένωσης είναι παραμελημένες. Ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η εδαφική συνεργασία της Ένωσης είναι απτό εργαλείο ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των περιφερειών που διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και βοηθούν τις περιφέρειες να λύσουν κοινά προβλήματα. Επίσης, η ενίσχυση ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ πόλεων και ε, βοηθά την ε, ανάπτυξη της αστικής πολιτικής. Μην ξεχνάτε ωστόσο ότι η εδαφική συνεργασία στην Ένωση έχει να κάνει με τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της συνοχής και την βελτίωση της ε, ανάπτυξης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις όπως την εδαφική, ε, την ε, καινοτομία στην εδαφική συνοχή. Συμφωνούμε ότι προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ενίσχυση της ειρήνης στην περιοχή στο πλαίσιο και της διεύρυνσης και της πολιτικής γειτονίας αλλά και ανά τον κόσμο μέσω της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών. Η συνεργασία αυτή βοηθά τις περιοχές που βρίσκονται εντός και εκτός των εξωτερικών σύνορων να αποκτήσουν, να γίνουν ε, ισχυρή οικονομική πόλη. Περισσότερα πράγματα θα προκύψουν από τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Ευχαριστώ. Ο κύρι, η κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από το 7 ως το 13 χρηματοδοτεί προτίθηκαν 8.000 έργα ε, συνοριακής ε, συνεργασίας σε περιοχές της Ευρώπης, εντός και εκτός της Ένωσης. Τα περισσότερα αφορούσαν 60 διασυνοριακές ε, περιοχές στην Ένωση και οι πολίτες που ζούσαν σε αυτά είχαν ναι μεν μικρό προπολογισμό αλλά με πολλά και θετικά αποτελέσματα υπήρξε πρόοδος στην ασφάλεια, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην κατάρτιση και βεβαίως δημιουργήθηκαν και θέσεις εργασία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο, προγραμματική περίοδο 14-20, ιδίω αν λάβουμε υπόψη τις ε, προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρέχει το φαινόμενο της μετανάστευσης. Ε, πρέπει να δοθεί σημαντικότερος ρόλος στις ανανεώσιμες ενέργειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στις περιοχές αυτές. Δεν πρέπει να μην συμφωνήσουμε με κάποιες πτυχές από την έκθεσή σας, ιδίως ό,τι αφορά την καθυστερημένη υιοθέτηση των προγραμμάτων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις στη νέα στη νέα προγραμματική περίοδο. Συμφωνούμε επίσης το ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα διασυνοριακά δεδομένα. Και εμείς ε, ζητούμε όπως και εσείς από την Επιτροπή και την Eurostat να μας δώσει αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να είναι είμαστε πιο προσεκτικοί στην χρήση κάποιων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προτείνει η συγγήτρια. Οι δύο, δύο παραγράφους, τις 23, την 23 και την 28, το έχουμε πει άλλωστε και σε άλλες ευκαιρίες, ότι δεν εγκρίθηκε, δεν διαπιστώθηκε μάλλον ότι τα εργαλεία αυτά έχουν προσθέμενη αξία στις πολιτικές συνοχής, γιατί επιπλέον ε, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς πολύ, ε, πολύ ε, εμπλεκόμενοι. Θα φύγω γιατί δεν θα δηλαδή, είχα καθυστερήσει και πρέπει να φύγω γιατί νόμιζα θα τελειώναμε νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χουαρίστη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εν συντομία, κυρία Πρόεδρε, να σχολιάσω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματικούς ε, στόχους, ε, προτεραιότητες για να μην είναι περιοριστική και να προσαρμοστεί καλύτερα στις διαφορετικές πραγματικότητες. Επίσης, η οδαφική συνεργασία δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στα διασυνοριακά προγράμματα μικρότερης κλίμακας πρόταση απλούστευσης θεωρώ ότι θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη, διότι ο κανονισμός έχει πολλές απαιτήσει και είναι άκρος πολύπλοκος για αυτά τα project. Επίσης, καμία δαυκή συνεργασία δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν είναι εγγυημένη συμμετοχή των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών και αυτό από την πρώτη στιγμή. Χρειαζόμαστε πιο σαφή καθοδήγηση και κατευθύνηση ως προς αυτό σε ό,τι δεν αφορά την αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών και δύο τελευταίες ανησυχίες, οι φυσικά είναι μια γενική αρχή πολύ καλή, όμως όχι αν συνεπάγεται ότι η πολιτική συνοχή τελικά θα γίνει ε, ένα είδος ε, ε, μικρού εύση. Και θα πρέπει να δούμε με το μικροσκόπιο τη συμπράξη δημοσιοδητικού τομέα, διότι κάποιε εμπειρίε που έχουμε, παραδείγματο χάρη από το Ισπανικό κράτο, μα δείχνουν ότι υπήρξε κακοδιαχείριση τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάκοβτσιτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση. Σημαντικό είναι λοιπόν το ότι τονίζεται την σημασία της ε, εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Το Ίντερεγκ έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό ρόλο σε διάφορες ε, περιφέρειες της Ευρώπης και αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε βέβαια αυτό το πρόγραμμα και τις νέες διαστάσεις που έχει. Μία από αυτές είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν μακροπεριφέρειες. Εγώ είμαι εισηγητής για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Έχουμε και την μακροπεριφέρεια των Άλπαιων και άλλες πρωτοβουλίες. Βλέπω λοιπόν διάφορες λύσεις αλλά και προβλήματα. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, γιατί πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Συχνά θέλουν οι τοπικές αρχές στις δύο πλευρές των συνόρων να χρηματοδοτήσουν παραδείγματο χάρη ένα σιδηροδρομικό έργο ή έναν αυτοκινητόδρομο και τα κράτη μετά δεν θέλουν να βρουν τέτοιες λύσεις ή να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο ή και το αντίστροφο μπορεί να σημαίνει Αυτό το οποίο θέλω να πω εν πάση περιπτώσει είναι ότι έχουμε πολλούς μηχανισμούς που αναπτύσσονται και κάστον δυνατά τα μεγάλα και μικρά διασυνοριακά έργα. μέσω του Ίντερεγ ή άλλων περιφερειακών έργων. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις για να ενισχύσουμε πραγματικά την εδαφική συνεργασία και την διασυνοριακή συνεργασία. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κοινή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ και Χωρίς μικρόφωνο. Mm Τώρα δουλεύει. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας κύριε Πρόεδρε, έκθεση η οποία καλύπτει όλες τις ε, πτυχές της ε, εδαφικής συνεργασίας και έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς εδώ και χρόνια προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα, γιατί πάντα την πληρώνουν οι μεθοριακές ε, περιοχές, οι οποίες ανήκουν στις πιο αδύναμες ε, περιοχές ε, και ειδικά εκεί όπου έχουμε εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει πλέον έκτημα. Έχουμε λοιπόν το μέσο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και Αναφέρατε βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον σύνδεσμο για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ως ένα νομικό μέσο και πράγματι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διασυνοριακή συνεργασία στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, κάτι το οποίο βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε και από τις ειδήσει και τον τύπο ότι κάθε μέρα θα είναι όλο και πιο σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν πως η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ δύο περιφερειών μεθοριακών είναι κάτι το οποίο παρακολουθούν πάντα οι κεντρικές αρχές με καχυποψία, φοβούνται για την κυριαρχία τους, ε, πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε και να δημιουργήσουμε τη βάση έτσι ώστε οι μεθοριακές περιοχές να ε, συνεργάζονται καλύτερα και να έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες και ελπίζω η έκθεση αυτή να συνεισφέρει σε αυτό. Αναφέρεται επίσης πως ε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την καλύτερη νομοθεσία για τη διασυνοριακή συνεργασία Βεβαίω τώρα έχουμε πια Ολλανδική Προεδρία και ελπίζω και η Προεδρία αυτή να ακολουθήσει την προσέγγιση του Λουξεμβούργου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει τον λόγο. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Άγνες τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζουμε την έκθεση. Συμφωνούμε απόλυτα με την προστιθέμενη αξία της συνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη. Όπως και η πρόεδρος, πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη, όχι μόνο γιατί θα επηρεάσει την ενδιάμεση να θεωρήσει ο δεύτερος στόχος, όπως ξέρετε, της συνοχής, την εδαφική συνεργασία το Ίντερεγκ δεν εμπλέκεται από την ενδιάμεση αναθεώρηση όπως βάση του κανονισμού για, ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά για την προετοιμασία κυρίως στοιχείων προς επίδοση των αλλαγών στο επόμενο, ε, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ως προς την σύσταση 37 δεν έχουμε θέση για τον προπολογισμό που πρέπει να δοθεί, αλλά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε όπως κάναμε και στις πρώτες συζητήσει στο τέλος του 15 σε ό,τι αφορά την διανομή, πληρώσαμε μεγαλύτερη προσοχή στις δεσμεύσεις που κάναμε το 2011 για μια δίκη διαμονή μια, μια δίκαιη διανομή των αναγκών. Κάνουμε τώρα μια μελέτη που έχουμε αναθέσει για τις ανάγκες των συνόρων που θεωρούνται ως εμπόδια και ταυτόχρονα δυνατότητα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι δύσκολο διότι όπως είπατε ο στόχος μας είναι να έχουμε έναν στόχο όσο πιο επιστημονικό γίνεται για να δημιουργήσουμε ε, τις δυνατότητες να έχουν οι νομοθέτες ε, στρατηγικές για τα σύνορα. Αυτό είναι το πλάνο και μπορούμε να σας ενημερώσουμε προς το τέλος του έτους όταν ετοιμαστούν οι μελέτες. Με βάση την εμπειρία μας μπορούμε να σας πούμε ότι όντως η συνοριακή συνεργασία δεν είναι εύκολη και μια ενδιάμεση, ένα ενδιάμεσο επίπεδο δεν θα είναι αναγκαστικά θετικό. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση 41 και την πρόταση του, της Λουξεμβουρκιανής Προεδρίας, μια άλλη μελέτη που ξεκίνησε η Επίτροπος Κρέτου πριν, πέρυσι, πρόπερση, βρισκόμαστε στην, είναι σε δύο επίπεδα, βρισκόμαστε στη φάση, στην πρώτη φάση, την εντοπισμό των εμποδίων και το δεύτερο, το διαπιστώνει ωστόσο ότι το πρώτο εμπόδιο είναι η κινητικότητα των εργαζομένων. Η διαβούλευση που κάναμε για τρεις μήνες επίσης αυτό έδειξε. Η δεύτερη φάση είναι πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα εμπόδια, ποιες είναι οι βέλτιζες πρακτικές, οι εναλλαγικές λύσεις και η πρόταση του Λουξεμβούργου θα είναι μία από τις προφανώς σοβαρές εναλλακτικές. Η Επιτροπή έχει πρόθεση να παρουσιάσει ένα κείμενο με τα βασικά θέματα στις αρχές του 17. Σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι η προσέγγιση κομισιών αυτή που χρειαζόμαστε, αλλά μια πολυεπίπεδη. Τώρα, για το θέμα της ορατότητας των επιτευγμάτων του Ίντερεγκ. με χαρά μπορώ να σας πω ότι ο προϋπολογισμός στηρίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων και Υπάρχουν πάρα πολλά project του Interreg. Χρησιμοποιήστε τον, το χάρτη αυτό, γιατί είναι ένας χάρτης, για να δείτε στη συγκεκριμένη εκλογική σας περιφέρεια τι έχουμε πετύχει. Αυτό είχε ζητήσει η Αντιπρόεδρος Γεωργίευα. Εμείς το τροφοδοτούμε συνεχώς για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα που είδαμε ήταν ε, το πρόγραμμα ε, αποναρκοθέτησης ε, μεταξύ Ουγγαρίας και Κροατίας. Η μεγάλη περιφέρεια των Grand Region είναι ένα παράδειγμα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Αυτός ο χάρτης είναι χρήσιμος, χρησιμοποιήστε τον. Νομίζω ότι κάλυψα τα πάντα. Ε, ε, μία παρέμβαση νομίζω θέλει κάποια διευκρίνηση για τη μετανάστευση. Η κυρία Κρέτσου ζήτησε από τα κράτη-μέλη, εμείς ζητάμε από τα προγράμματα, να χρησιμοποιούν τα ταμεία όσα έχουν με το μενού που έχουμε στη διάθεσή μας. Τους 11 θεματικούς στόχους δηλαδή για να ενισχύσουμε την ένταξη των μεταναστών, τρεις θεματικοί στόχοι έχουν εντοπιστεί ως ε, πιθανό να βοηθήσουν μετανάστες, 8, 9 και 10. Για τα, ιδίως για το Interreg έχουμε τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων για άμεσα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν. Κάποια προγράμματα ήδη έχουν ξεκινήσει δράση στον τομέα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να παράσχουμε συγκεκριμένα project γρήγορα. Αλλά συνεχίζεται, συνεχίζονται οι προσκλήσεις για να βοηθήσουμε την ένταξη των μεταναστών. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα σχόλια και την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή και τις συστάσεις σας. Περιμένω και τις τροπολογίες. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία. Τετάρτη 6 Απριλίου για την κατάσταση των τροπολογιών. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο της διάταξης. Προφορική ερώτηση με ψήφισμα Η κυρία Μάλετη, εκ μέρου του ΕΛΚ, έχει κάνει την σχετική πρόταση για την επιτάχυνση τη υλοποίησης τη πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να σα θυμίσω ότι το ερώτημα, αυτή η προφορική ερώτηση, υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 128 του κανονισμού και αποφασίσαμε από κοινού με τους συντονιστές και με βάση τους ειδικούς κανόνες της Επιτροπής ΡΕΓΚΙ να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με την προφορική ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματος και να δούμε στο μέλλον πώς θα προχωρούμε γιατί αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Η κυρία Μάλιτιτς έχει τώρα το λόγο για να μας παρουσιάσει τις ιδέες της για την προφορική αυτή ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που υποστήριξαν τις ε, ερωτήσεις μου γιατί ήδη συζητήσαμε κάποιες ερωτήσεις που προτάθηκαν και τώρα έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω πως ε, το ψήφισμα αυτό και το θέμα γενικά η, η επιτάχυνση της εφαρμογής πολιτικής συνοχής είναι κάτι το κατεπήγον αυτή τη στιγμή γιατί βασικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμογή και οπωσδήποτε έτσι θα χάσουμε κονδύλια στο τέλος του 2017 και 2018 γιατί εφαρμόζουμε τον κανόνα νη συν 3 στην πολιτική συνοχή 14-20. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Ξέρω πως μπορεί κάποιος ε, να διαφωνήσει μαζί μου και να ρωτήσει χρειάζονται βοήθεια και γιατί δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως. Αλλά αν ε, αναλύσουμε το τι εισάγεται εδώ πέρα με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 βλέπουμε πως έχουμε πολλές καινοτομίες για τα κράτη-μέλη και δεν, ε, είχαμε, δεν είχαν τόσο ε, καιρό για να προετοιμαστούν γιατί υπήρχε η δεματική εστίαση, εστίαση στα αποτελέσματα, συντονισμός με την οικονομική πολιτική, προτεραιότητες της Ένωσης και περιφερειακές ανάγκες, πιο συντονισμένη χρήση των κονδυλίων, οπότε για να τα υπάρχουν όλα αυτά, όλα αυτά στην πράξη έγιναν με έναν τρόπο ώστε εγκρίθηκαν πολύ αργά τέλος του 2014 τα επιχειρησιακά προγράμματα και τώρα όταν κοιτάμε την εφαρμογή και το που είμαστε με την εφαρμογή σε πολλά κράτη-μέλη δεν έχουμε καθόλου έργα που να έχουν δοθεί σε αναδόχους μόνο 0,5% των ε, κονδυλίων ε, που αναλογούν στο πρώτο έτος. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια περισσότερα μέτρα. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από την Κομισιόν με το ψήφισμα αυτό να προετοιμάσει μια λεπτομερή ανάλυση για τους κινδύνους αποδέσμευσης ποσών στα κράτη-μέλη. Θεωρώ πως σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε εγκαίρως και πρέπει πράγματι να συνεχίσουμε με την ομάδα συνεργασίας που είχε ξεκινήσει την περίοδο 2007-2013 αλλά τη χρειαζόμαστε και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και θα θέλαμε οπωσδήποτε η Κομισιόν να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης ε, των δραστηριοτήτων της Τασκός ε, ανά κράτος μέλος. Επίσης να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις δράσεις που προβλέπονται για να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για εφαρμογή και αξιολόγηση γιατί η διοικητική ικανότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την έγκυρη εφαρμογή και μετά βεβαίως να επιταχυνθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την απλοποίηση. Γνωρίζουμε πως έχουμε το σχέδιο δράσης το οποίο τελειώνει το 2019 και είναι πολύ αργά και επίσης θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει για τα μέτρα τα οποία προβλέπει για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2016. Αυτό αφορά τα έργα τα οποία ακόμα έχουν συσσωρευτεί και βεβαίως τώρα μειώνονται αυτά αλλά θα αυξηθούν ξανά στο μέλλον γιατί τι γίνεται έτσι χάνουμε την αξιοπιστία μας στην πολιτική συνοχής. Επίσης να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και πράγματι να δούμε τι γίνεται και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τελευταία ερώτηση προς την Κομισιόν. θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων με τεχνικούς ε, και οικονομικούς όρους για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των έργων γιατί σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς και δεν έχουν τα κράτη τη δυνατότητα να προετοιμαστούν ε, και μετά να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι ένα καλό μέσο για να στηρίξει και να βοηθήσει. Το λέμε, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να έχουμε κάποια συγκεκριμένα τέτοια σχέδια. Τέλος, στόχος είναι να έχουμε μια συζήτηση για όλες αυτές τις πληροφορίες από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε μετά με βάση αυτά να μπορούμε να δούμε εάν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι στον κανονισμό γιατί εισάγονται τελείως νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής στον κανονισμό 2014-20 και ίσως χρειάζεται λίγη περισσότερη ευελιξία για να βοηθήσουμε να στηρίξουμε τις χώρες για να εφαρμόζουν εγκαίρως τα πράγματα και να επιτυγχάνουν κάποια αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχετε στο φάκελό σας την πρόταση ψηφίσματος. Ακούσατε την κυρία Μάλετιτς. Σας έκανε μια αναλυτική παρουσίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και 12 το μεσημέρι χρόνο για να υποβάλουμε τροπολογίες εφόσον το επιθυμούμε ώστε η ψηφοφορία να γίνει τον Απρίλιο και η συζήτηση, μάλλον θα υποβάλουμε και αίτημα για την ολομέλεια στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε συζήτηση, χρειαζόμαστε κύριε Φανίστελ μία παρατήρηση. Μάλιστα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θα κάνουμε τις τροπολογίες μας, αλλά Έχουμε αυτή τη διαδικασία με τις ε, προφορικές ερωτήσεις για να ε, συζητάμε και στην Ολομέλεια κάποια θέματα. Νομίζω ότι στόχος είναι να έχουμε μια κοινή συζήτηση το Μάη στην Ολομέλεια. Ξέρετε, υπάρχει πολιτική, αλλά αν ε, βάλουμε το χέρι στην πληγή, είναι να δούμε τι έγινε την προηγούμενη περίοδο 7-14 και τις μη εκμεταλλευστήσεις πιστώσεις. 3 με 9 δις είναι το ποσό που εκτιμάται ότι θα γυρίσει πίσω τα ταμεία των κρατών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο των τύπων των ύλων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορώ να τα διαβάσω αλλά δεν νομίζω ότι η διατύπωση είναι αρκετά ισχυρή. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε πριν την ψηφοφορία να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση. Γιατί εδώ το θέμα που τίθεται είναι γιατί θέλουμε αυτή την προσφορική ερώτηση, θέλουμε να επηρεάσουμε. Επειδή είπατε ότι θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να σχέδιο δράσης από την Κομισιόν για την Ιταλία. Μας τα είπαν και πριν. Γιατί μισή Ιταλία δεν υπάρχουν σχέδια. Θα είναι τρομερό με τον ίσιν 3. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί υποβάλλουμε αυτή την προφορική ερώτηση. Που την υποβάλλουμε γιατί θέλουμε επιτάχυνση τώρα. Όχι να επιταχύνουμε τώρα, αλλά να συζητήσουμε μισή χρονιά, μετά από μισό χρόνο που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τα πράγματα με αυτή τη διαδικασία και όχι όταν υποβάλαμε τι ερωτήσει απευθεία στην Ολομέλεια. Ναι, λέει πρόεδρο, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Θέλετε να πείτε κι εσεί κάτι. Attenzione a come facciamo questo dibattito. Lo dico con, eh, con la serietà diciamo, del, del tema. Κοιτάξτε, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, Άμα είναι να συζητάμε για κάθε χώρα να συζητάμε, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε αλλιώς για την Ιταλία. Αν είναι να γίνει μια συζήτηση όπως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση για τους κινδύνους που είχαμε και για τη μελλοντική διοίκηση, ναι, τότε αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Χρειαζόμαστε επίσης να δούμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα μέσα που έχουμε π.χ. την Task Force ή αν θα συζητήσουμε το θέμα των διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων. Έτσι θα αποφύγουμε το να παγιθεύσουμε το σύμφωνο σταθερότητας ε, και αυτά τα θέματα στην πολιτική της ε, σύνοχης. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη στιγμή αυτή την συζήτηση. Πρέπει όμως να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Τι μιλάμε, για μεμονωμένες χώρες να μιλήσουμε για μεμονωμένες χώρες. Αν από την άλλη πρέπει να έχουμε μια συζήτηση η οποία θα βάλει στο κέντρο της, την Κομισιόν, εντάξει τότε αυτό είναι άλλο θέμα. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Αυτός είναι και ο σκοπός του όλου εγχειρήματο με τις τροπολογίες για το ψήφισμα και την προφορική ερώτηση, γιατί θέλουμε να καλύψουμε όλες τις ε, απόψεις και να ε, δημιουργήσουμε μια κοινή θέση που θα μας αντιπροσωπεύει. Σε Επιτροπή Δευτέρα, 21 Μαρτίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Και θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Απρίλιο και μάλλον τον Μάιο στην Ολομέλεια. Αυτά για αυτό το σημείο. Και εδώ λίγη η δημόσια συνεδρίαση και συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Να παρακαλέσω τα μέλη της Επιτροπής που δεν είναι συντονιστές να αποχωρήσουν, γιατί δεν μας μένουν παρά 25 λεπτά.